Eh, Θα ήθελα να καλωσορίσω τους συναδέλφους και τους παρευρισκόμενους στη σημερινή συνεδρίαση και τους διερμηνείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίσατε λοιπόν όλοι στη σημερινή μας συνεδρίαση. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον απόγευμα. Το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση των πρακτικών. Η έγκριση της ημερήσιας διάταξης, συγγνώμη. Έχουν γίνει κάποιες μικρές αλλαγές το σημείο 5 και το σημείο 6, δηλαδή οι προφορικές ερωτήσεις και το ψήφισμα για τη βία, θα συζητηθούν από κοινού, τα σημεία 5 και 6 από κοινού. Για τα 7 και 8 ακριβώς το ίδιο, θα τα εξετάσουμε από κοινού. Και θα συζητήσουμε αύριο, μετά το 10 μετά το σημείο 10. Το σημείο 11, το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, αύριο θα συζητηθεί στις 11. Αυτές οι μικρές αλλαγές έγιναν. Μπορείτε να εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Ναι, ωραία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης που έγινε την 1η Σεπτεμβρίου έχουν κυκλοφορήσει δεν είχαν ε, υποβληθεί κάποιες παρατηρήσεις για τα πρακτικά μέχρι να η σημερινή συνεδρίαση, οπότε κρίνω ότι εκρίνονται και τα πρακτικά. Οι ανακοινώσει Προέδρου τώρα, σημείο 3. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η Έλληνα Μανιάτη από την Γραμματεία θα φύγει από 1η Οκτωβρίου γιατί θα πάει στην Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών. Εξ ονόματος ολόκληρης Επιτροπής μας θέλω να ευχαριστήσω την ε, Ελένα ε, για, τις, για τη δουλειά της και πραγματικά καλή τύχη σου ευχόμαστε. Τα μέλη της Επιτροπής μας τώρα θα προσκληθούν σε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Στις 12 Οκτωβρίου θα γίνει κοινή συνεδρίαση, 6 με 7. Ε, ο δόκτωρ Άσαφος Μιγκύρο, που είναι ο Γενικός Γραμματέας ε, του των Ηνωμένων Εθνών θα παρευρεθεί και φυσικά ε, σας καλωσορίζουμε όσοι θέλετε να έρθετε, είστε ευπρόσδεκτοι και θα σας ε, ενημερώσουμε με την μερίσια διάταξη, το χώρο και τη συνεδρίαση, την αίθουσα δηλαδή της συνεδρίασης. Ελπίζουμε να ε, υπάρξει αθρό προσέλευση σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Αυτά για τα τρία πρώτα σημεία και πάμε στο σημείο 4. Μας έχει ανατεθεί εντολή να ορίσουμε ε, να ορίσουμε υποψηφίους για το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Ε, και ναι, θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερη τιμή που μας ανατέθηκε αυτή η εντολή. Οι συντονιστές έχουν ε, νωρίτερα αποφασίσει για την ε, μέθοδο εργασίας που θα ακολουθήσουμε για τον ορισμό των υποψηφίων. Όλα τα μέλη είχαν την δυνατότητα να προτείνουν υποψηφίους για το φόρουμ εμπειρογνωμόνων και λάβαμε διάφορες προτάσεις. Την 1η Σεπτεμβρίου αποφάσισαν λοιπόν οι συντονιστές ότι θα ορίσουμε έξι ε, υποψηφίους που θα προσκαλούσαμε στη συνέχεια στην Επιτροπή μας. Σε αυτό το στάδιο είμαστε σήμερα, τους έχουμε προσκαλέσει και έχουμε λάβει πληροφορίες για τις έξι υποψηφίους, για την εμπειρία τους στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων και θα μας εξηγήσουν ε, τι κατά τη γνώμη τους μπορούν να συνεισφέρουν ε, στο φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Έξι υποψηφίους έχουμε σήμερα, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί τους. Κάθε υποψήφιος θα ε, μιλήσει 10 λεπτά για να μας εξηγήσει ποια εμπειρία έχει, στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων και τι μπορεί να προσφέρει στον τομέα. Μετά θα έχετε τη δυνατότητα ε, για 10 λεπτά να θέσετε ερωτήσεις. Θα πάρουμε με τη σειρά όλες τις ε, προτινόμενες υποψηφίους και αύριο οι συντονιστές ε, θα αποφασίσουν ε, για τον διορισμό ανάμεσα σε αυτές τις έξι υποψηφίους που θα συναντήσουμε σήμερα. Αυτή θα είναι η μέθοδος μας για το σημείο αυτό της μέσης διάταξης. κάλος ορίζω την πρώτη υποψήφια για το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων, η κυρία Λίζε Κέλλη, που είναι διευθυντής στην μονάδα μελετών για την κακοποίηση παιδιών και γυναικών ε, στο Πανεπιστήμιο London Metropolitan. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος που ήρθατε σήμερα. Καλωσορίσατε κυρία Λίσκελη ε, στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο για περίπου 10 λεπτά. Aha, Okay. Thank you, Madam um, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που μου δίνετε να ε, θέσω την υποψηφιότητά μου ως μέλος ε, του, της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ε, στο σύντομο χρονικό διάστημα που έχω στη διάθεσή μου θα σας πω λίγα πράγματα για το παρελθόν μου και για το πώς θεωρώ ότι το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των θεμάτων που αφορούν στην ισότητα των γυναικών. Μας ενδιαφέρουν οι δράσεις ε, προτεραιότητας, έχουμε το πρόγραμμα Δάφνη και υπήρχε και ένας μειοδοτικός διαγωνισμός ε, για την εναρμόνιση της ε, νομοθεσίας. Οι μελλοντικέ δράσεις του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Γενικών θα είναι σημεία αναφοράς για το Ινστιτούτο για τα θέματα ισότητας των φύλων. Εγώ ασχολούμαι με τα θέματα αυτά για πάνω από 30 χρόνια ως ακαδημαϊκός, ως ε, ε, άνθρωπος του χώρου και θεωρούμε πλέον εμπειρογνώμων ε, σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Πέρσι εργάστηκα σε ένα πρόγραμμα για τους δείκτες και για τους ελάχιστους, ελάχιστες προδιαγραφές για τα θέματα φύλου. Ε, με ενδιαφέρουν διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών, ε, η βία στο σπίτι, η σεξουαλική βία, διακίνηση ανθρώπων ε, και διάφορες άλλες πρακτικές βίας. Όπως επίσης και θέματα κακοποίησης παιδιών και προστασίας παιδιών. Το κέντρο με το οποίο συνεργάζομαι έχει περατώσει πάνω από 100 προγράμματα και διεθνή και εθνικά. Με το πρόγραμμα Δάφνη ε, ετοιμάσαμε μία μελέτη, μία αναφορά και πολλές ε, υποθέσεις ανά την Ευρώπη και είχα το χαρά να συνεργαστούμε πολλούς ε, ακαδημαϊκούς ανά την Ευρώπη. Έχουμε θεσπίσει συγκεκριμένε μεθέδου και έχουμε φήμη ότι καθορίζουμε συγκεκριμένε πολιτικέ οι οποίε μπορούν να βοηθήσουν σε θέματα νομοθεσία, πολιτική και πρακτικών. Και αυτό για μένα είναι ε, το τεστ, ε, το κατά πόσον η δουλειά που κάνουμε κάνει τη διαφορά. Δεν έχουμε μόνο εικόνες, έχουμε και ένα μητρό κακοποίησης. Ε, η προστασία των γυναικών μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική αν έχουμε ταυτόχρονα και προστασία των παιδιών και Κάνουμε πολλές ε, εργασίες ε, στη χώρα μου με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, με το Υπουργείο Δικαιοσύνη και τις αστυνομικέ δυνάμεις. Ω Επίτροπος ε, για την Επιτροπή Γυναικών, την Εθνική Επιτροπή Γυναικών, συνεργάστηκα με πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οι οποίες δεν είχαν στο παρελθόν συνεργαστεί. Πλέον αναγνωριζόμαστε ω ένα πολύ σημαντικό εταίρος σε πολλού τομεί πολιτική. Έχουμε μελέτες για τις γυναίκες ε, από το 1988 και έχουμε πλέον το μόνο πρόγραμμα μάστερ στον κόσμο για κακοποίηση γυναικών και παιδιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όσους δραστηριοποιούνται στον χώρο να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις όχι μόνο σε θέματα θεωρίας ισότητας των φύλων αλλά και στην ε, πράξη. Για μένα όλα τα θέματα αφορούν τα θέματα των φύλων. Η ανάλυση των φύλων μας επιτρέπει να δούμε τι διαφοροποιημένες επιπτώσεις έχουμε σε γεγονότα και πολιτικές σε σχέση με τους άνδρες και τις γυναίκες και αυτό έχει και κάποιες έννοιες όπως είναι η ελάχιστη ασφάλεια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και φυσικά και η τρέχουσα οικονομική κρίση. Για να μπορέσουμε όμως να είμαστε αποτελεσματικοί θα πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς η ανάλυση της ε, σχέσης των φύλων και θα πρέπει να Βλέπουμε και τι γίνεται και από θεωρητικές σκοπιά ε, σε ακαδημαϊκά θέματα. Ε, πρόσφατα τέθηκε το θέμα της αναλογικότητας. Ένας από τους λόγους για του οποίου θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα Ινστιτούτο για θέματα φύλου είναι ότι δεν υπάρχει πλέον τόσο μεγάλη αρμοδιότητα ε, πολλοί από τους ανθρώπους που συναντώ θεωρούν ότι τα θέματα φύλου αφορούν μόνο γυναίκες, ενώ ε, έχει να κάνει και ε, η αλληλεπίδραση μεταξύ ανδρών και γυναικών που, διαφορετικών ηλικιών που επηρεάζονται από τα ίδια θέματα. Και επίσης έχουμε θέματα εφαρμογής καινοτόμων θεμάτων σε θέματα ισότητας φύλων και προσπαθούμε να δούμε ε, διάφορα θέματα που αφορούν ε, στα φύλλα ε, και πώς μπορούν να εντοχθούν αυτά στις πολιτικές για την ισότητα των φύλων. Ανάλογα με το δείγμα που έχουμε και τις μορφές βίας που διαπιστώνουμε σε κάποιες έρευνα, μεταξύ κάποιων ηλικιών οι γυναίκες έχουν υποστεί βία τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Και Υπάρχουν σχέσει σε θέματα ηλικία και αναπηρία. Για παράδειγμα, οι νεότερες γυναίκε γυναίκες είναι πιο ευάλωτε σε βία. Επίση, θα πρέπει να εξετάσουμε ει βάθο και τι συνέπειε τη βίας. Ε, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά τι γίνεται στις οικογενειακές και πιο στενές σχέσεις, αλλά μπορεί να έχουμε βία σε εργασιακούς χώρους, σε χώρους διαμονής, σε αθλητικούς χώρους και φυσικά και στα ε, θέματα που αφορούν στη μετανάστευση. Επίσης γνωρίζουμε ότι η επαναλαμβανόμενη βία, η οποία δεν αντιμετωπίζεται, έχει πολύ σημαντικές ε, συνέπειες και στην παιδεία και στην ε, συμμετοχή στα κοινά και στη δημόσια υγεία, στο να είναι κάποιος γονέας, στην κοινωνική συνοχή και στην κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτά λογικά θα πρέπει να αρκούν ω στοιχεία για να θέσουμε τη βία στο επίκεντρο, διότι ε, έχει να κάνει με όλα τα θέματα που άπτονται τη ισότητα των φύλων. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα λίγο. Υπάρχει περίπτωση η βία να είναι ε, μια συγκεκριμένη και σε, κάποιες, ε, σε κάποιο βαθμό ανεξάρτητη δομή που οδηγεί στη βία. Και αυτό σημαίνει ότι, στην ανισότητα, συγγνώμη, και αυτό σημαίνει ότι ε, μπορεί να μην προοδεύει. Η μείωση λοιπόν ε, της βίας δεν μπορεί να προβλεφθεί. Ε, μπορεί να υπάρχει, για παράδειγμα, μεγαλύτερη απασχόληση για τις γυναίκες, ίση μισθοδοσία. αυτά είναι τα παραδοσιακά στοιχεία που αναζητούμε για την ισότητα των φύλων και υπάρχει και μια θεωρία ότι ισχύει το αντίθετο, ότι η βία κατά των γυναικών μπορεί να προκύψει λόγω της μετάβασης προς την ισότητα των φύλων. Το παράδειγμα εδώ είναι οι σκανδιναβικές χώρες και πιο συγκεκριμένα η Σουηδία, όπου οι δείκτες ε, βίας κατά των γυναικών βρίσκονται στην, ε, σε πολύ ψηλά επίπεδα και εκεί φαίνεται ότι η ισότητα είναι πολύ μεγαλύτερη από κάποιες χώρες όπου οι αλλαγές είναι πολύ πιο βραδίες. Έχει πολύ μεγάλα ποσοστά η Σουηδία στην, ε, σε σχέση με την Ευρώπη, διπλάσια από αυτά του Ηνωμένου Βασιλείου και ε, τριπλάσια από αυτά της Γερμανίας. Εάν λοιπόν μία ε, έμεση συνέπεια της ισότητας των φύλων είναι η βία, είναι ε, κάτι το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε. Έχει αναγνωριστεί, αναγνωριστεί σε κάποιες μελέτες, αλλά θα πρέπει να το δούμε γενικότερα, να αναγνωριστεί παγκόσμια. Το κέντρο μας είχε μεγάλες επιπτώσεις σε θέματα ισότητας των φύλων, αλλά δεν έχει γίνει πολύ, πολύ μεγάλη πρόοδο σε θέματα βίας και διακίνησης ε, ε, συγχρόνου λαθρεμπορίου γυναικών. Επομένως θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, βία στο σπίτι, ε, διότι δεν θα πρέπει να παραμεληθούν και θα πρέπει ε, η Ευρώπη να θεωρηθεί ένα εργαστήριο στο οποίο δοκιμάζουμε διάφορες πολιτικές. Μπορούμε να μάθουμε πολλά και εμείς αλλά και οι άλλοι. Και ο τελικός λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι η βία θα πρέπει να είναι βασικός τομέας είναι διότι ε, αρκετές γυναίκες είναι πιο επιφυλακτικές στην Ευρώπη από τους άνδρες, αλλά οι γυναίκες πάντα ασχολούνται με τη βία. Το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι οι περισσότεροι θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εστιάσει σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Ως εμπειρογνώμων λοιπόν θα μπορέσω να προσφέρω πολύ σημαντική εργασιακή εμπειρία, πολλά στοιχεία για την πολιτική ε, της βίας κατά των γυναικών και φυσικά θα συνεργαστώ αγαστά με την Επιτροπή Γυναικών για να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά σας συμπεριλαμβάνεται στις πρόσφατες έρευνες και στις, στα ερευνητικά κέντρα και θα μπορούμε να ακολουθήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την Επιτροπή σε θέματα απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κυρία Κέλλη, σας ευχαριστούμε θερμά. Τώρα ακούμε τα μέλη της Επιτροπής, αν υπάρχουν ερωτήσεις προς την κυρία Κέλλη. Ε, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Μετά από αυτά που άκουσα, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχάς, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία, κυρίως στο θέμα της βίας. Τι θα κάνετε για να προχωρήσει ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πρώτα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν και τι δυσκολίες πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε και ποια θα είναι για σας οι προκλήσεις ε, για το μέλλον ενός τέτοιου Ευρωπαϊκού Κέντρου. Ε, στρέφομαι προς τη Λίζ. Ε, θα ήθελες να απαντήσεις στο ερώτημα. Νομίζω ότι μία από τις ε, μεγαλύτερες δυσκολίες είναι να καταλήξουμε σε συνένεση σχετικά με το τι σημαίνει η ισότητα των δύο φυλών. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά πλαίσια στην Ευρώπη για την ισότητα των ε, φύλων. Δηλαδή σε κάθε χώρα ακολουθούμε διαφορετική μέθοδο. Κάποια κράτη τονίζουν, δίνουν έμφαση σε διαφορετικές ε, κατευθύνσεις πολιτικής αν θέλετε. Οπότε ε, το πρώτο καθήκον που πρέπει να επιτελέσουμε είναι να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε συνέντευξη σχετικά με την έννοια της ισότητας των δύο φίλων ε, στα διάφορα αρμόδια Ινστιτούτα και μετά να δούμε ποιοι είναι οι φραγμοί, ποιες είναι οι προκλήσεις ε, που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να το πετύχουμε αυτό στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει μάλλον περιφερειακή ε, σκοπιά γιατί διαφέρουν οι προκλήσεις ανάλογα με την περιοχή της Ευρώπης για την οποία μιλάμε. Η ισότητα των δύο φύλων ε, συχνά ε, είναι κάπως, ε, δεν, δεν είναι κεντρικό σημείο των πολιτικών ενώ θα έπρεπε περιθωροποιείται από τις πολιτικές και παρότι θα έπρεπε δεν συμβαίνει αυτό στην πράξη οπότε πρέπει να βρούμε ε, τρόπους ούτως ώστε να μην μένει στο περιθώριο αυτό το θέμα, ε, να εντάσσεται πραγματικά στις πολιτικές μας. Ε, και αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου στην έλλειψη γνώσεων σχετικά με τι σημαίνει ισότητα των φύλων και επίσης δεν αναλύονται παρκώς τα θέματα διότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη τεχνογνωσία ε, ακόμη και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και κυρίως στα πλαίσια των εθνικών μηχανισμών. Σας ευχαριστούμε, η κυρία Κουρνέλ. Ευχαριστώ, ιδίως ε, για τις ε, γνώσεις σας για τη βία κατά των γυναικών η οποία είναι εντυπωσιακή. Εδώ αναφερόμαστε σε όλα τα θέματα ε, τα οποία έχουν σχέση με τις γυναίκες και την ισότητα μεταξύ τους σε 30 χρόνια λοιπόν πήρας ε, σε γενικά θέματα προφανώς ε, έχετε ασχοληθεί και με άλλους τομείς όπως οι γυναίκες στη λήψη των αποφάσεων. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι επ' αυτού διότι προφανώς οι γνώσεις σας είναι εντυπωσιακέ αποφάσισα να σας πω τι θα μπορούσα εγώ να προσφέρω ε, σαν εμπειρογνώμων. Έχω ε, όμως ε, γνώση στον τομέα αυτό. Έχω υπάρξει επίτροπος στην Εθνική Επιτροπή για τις Γυναίκες και έχω ασχοληθεί με όλα τα θέματα για να μπορέσουν οι γυναίκες να συμμετάσχουν ε, ιδίως ε, διότι είναι μεγάλο βήμα για τις περισσότερες γυναίκες να προχωρήσουν έτσι και γι' αυτό αποφασίσαμε να επιτρέψουμε στις γυναίκες ε, να μπορέσουν να επέμβουν και σε τοπικό επίπεδο πράγμα το οποίο στοχεύει εις ε, το να έχουν σχέση με τις γυναίκες που βρίσκονται σε δημόσιους οργανισμούς. Ε, και στους καταλόγους είδαμε ότι οι γυναίκες αυξήθηκαν κατά πολύ στους καταλόγους και εφόσον ε, έχουν την εμπειρία μπορούν πολύ πιο εύκολα να έχουν πρόσβαση σε θέσεις αυτού του είδους και επίσης, ε, ε, επίσης ε, για τα θέματα ισότητος των φύλων όπου είναι κάτι το οποίο δίδει μεγάλη, μεγάλη ευθύνη σε πολλούς οργανισμούς και όπου είναι εύκολο να υπάρχει ένα πρόγραμμα ισότητος μεταξύ των φύλων και για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει να υπάρχουν οργανώσεις σε διάφορους τομείς και να καταρτίζουν στόχους τους οποίους θα επιτύχουν εντός μίας τριετίας. Στις πρώτες φάσεις καταφέραμε να αντιμετωπίσουν τις γυναίκες πολύ πιο σοβαρά από ό,τι στο παρελθόν. Η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να κάνω μία ακόμη ερώτηση. Τι πιστεύετε ότι θα είναι το μέλλον ε, χρειαζόμαστε νέα στρατηγική, περισσότερη ε, νομοθεσία, καλύτερη εφαρμογή, καλύτερο περιβάλλον για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε λύσεις. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο βασικό σημείο το οποίο θα μπορέσετε να επηρεάσετε με αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να σας πω ή το ένα ή το άλλο, διότι ε, θα πρέπει να έχουμε πολλές στρατηγικές και όχι μόνο μία. Αλλά θα πρέπει να επιτρέψουμε στους ανθρώπους να μπορέσουν να κινηθούν επικοδομητικά και όχι μόνο σε επίπεδο γυναικών για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με κρίση και σαν άντρες ε, και τα, τον ακαδημαϊκό χώρο ε, διότι ε, γιατί δεν ρωτούν ποτέ τους άντρες γιατί όλα τα εγκλήματα συνήθως έχουν διαπραχθεί από άντρες πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μειώσουμε την εγκληματικότητα και νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει καλύτερα από τις γυναίκες. Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέπτεστε και τρόπο ε, θέσεως των ερωτημάτων για να αλλάξουν οι στρατηγικές. Δεν νομίζω όμως ότι μπορώ να σας πω, μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι έχουμε μία στρατηγική και αυτή είναι και θα μας οδηγήσει εκεί που θέλουμε. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει τέτοια λύση. Υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν επέτυχαν αλλά που επέτυχαν μερικώς και πρέπει συνέχεια να κοιτάμε και να ψάχνουμε να βρούμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ήθελα και εγώ ίδια να κάνω ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Αρχικά ένα σχόλιο για την βία κατά των γυναικών. Σε κάποια κράτη βλέπουμε τα στατιστικά στοιχεία για τις καταγγελίες ε, για εγκλήματα βίας κατά των γυναικών. Είναι ε, ε, υψηλότερα σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Μας είπατε για τη Σουηδία ότι είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά. Και θέλω να κάνω μία ερώτηση. Εντάξει, είναι συνάρτηση της εθνικής νομοθεσίας σχετικά περί υποβολής καταγγελιών. Δηλαδή υπάρχουν περισσότερες καταγγελίες ανάλογα με την εθνική νομοθεσία, ανάλογα με την υποστήριξη που προσφέρεται ε, για τέτοιες σχέσεις ε, όπου υπάρχει μεγάλη βία. Και ε, επειδή έχεις μακρά εμπειρία στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση, να κάνεις ένα σχόλιο, να μας πεις ε, για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητα των Δύο Φύλων και το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων συγκεκριμένα κατά την κρίση σου, ε, πού θα έπρεπε να αποδώσουν προτεραιότητα, σε, ποιο, σε ποια ακριβώς ε, δράση. Τώρα, για τα δικαιώματα υποβολής Ε, αναφορών. Είναι ένα πράγμα που ε, απασχολεί πολύ τους εμπειρογνώμονες. Ε, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το ένα θέμα είναι κατά πόσο η αστυνομία και η εισαγγελία καταγράφουν με ακρίβεια τις καταγγελίες. Δεν αναφέρουν όλα τα στοιχεία που φτάνουν μέχρι αυτούς, αλλά σε κάποια κράτη υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με άλλες. Τώρα, ε, ε, μιλήσατε για την εθνική νομοθεσία. Δίκιο έχετε. Αν ε, ο ορισμός του βιασμού είναι ευρύ σε παραδείγματος χάρη, θα υπάρχουν περισσότερα εγκλήματα που θα εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Ε, το έχουμε εξετάσει αυτό το θέμα στη μελέτη και δεν εξηγούνται επακριβώς οι διαφορέ ε, που διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Μετά υπάρχει και η βούληση υποβολή αναφόρων, ε, καταγγελιών μάλλον, ε, από τα ίδια τα θύματα. Ναι, είναι θέμα διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Υπάρχει, σχετίζεται αυτό με το αν το κίνημα των γυναικών στη συγκεκριμένη χώρα έχει γύρει το ζήτημα, αν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό το θέμα ή αν οι ίδιες οι αρχές επιβολής του νόμου ξεκαθαρίζουν ότι καλωσορίζουν γνωρίζουν τέτοιε καταγγελίε. Και υπάρχει και κάτι άλλο στο οποίο δεν μπορούμε να απαντήσουμε αν υπάρχουν διαφορετικά δηλαδή επίπεδα βία ανάλογα με τη χώρα και διάφορα είδη βία ανάλογα με τις χώρες. Ε, προσπαθήσαμε, ε, έγιναν απόπειρες να πούμε ότι όχι, είναι ε, ίδια η κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη, αλλά νομίζω εγώ ότι είναι πολύ πιο περίπλοκο το ζήτημα. Δεν μπορούμε να εξομοιώσουμε τις καταστάσεις, αλλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι ισχύει. Για τις προτεραιότητες τώρα που με ρωτήσατε για το Ινστιτούτο, ε, κατά τη γνώμη μου, η προτεραιότητα, δύο προτεραιότητες πρέπει να υπάρχουν. Πρώτον, η θεσμική φραγμή για την ε, αντιμετώπιση των θεμάτων ισότητας των δύο φύλων ε, και να έχουμε ένα ευρύ φάσμα δράσεων για να ενταχθεί το ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων στι γενικότερες πολιτικές, είτε μιλάμε για τα εθνικά κοινοβούλια, είτε μιλάμε για ε, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή πρέπει να ανανεωθεί η δέσμευση που έχουμε αναλάβει για την προώθηση της ε, ισότητας, γιατί υπάρχουν κάποιοι που δεν το έχουν αναδείξει σε προτεραιότητα αυτό το θέμα. Τώρα, η άλλη διάσταση του ζητήματος είναι να δούμε, να εντοπίσουμε τις βασικές προκλήσεις για τις ίδιες τις γυναίκες ε, βράχει πρόθεσμα και ε, ε, μέσο πρόθεσμα και να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτά. Ευχαριστούμε. Έχουμε άλλες δύο ερωτήσεις. Ο κύριος Σιμάνσκι και η κυρία Κώστα. Ο κύριος Σιμάνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ακούσαμε από εσά. Σας είμαι ευγνώμων που ασχοληθήκατε με το θέμα της αρενοπότητας και είπατε ότι το θέμα δεν έχει να κάνει μόνο με τις γυναίκες αλλά και με τους άνδρες. Και αυτό αποδεικνύει ότι πρόκειται για επιτροπή ίσων δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και ε, γυναικών. Δεν ξέρω βέβαια αν το Κοινοβούλιο θα έχει ποτέ επιτροπή δικαιωμάτων των ανδρών, αλλά ε, τέλος πάντων τα πράγματα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Έχω μια πρακτική ερώτηση να σας κάνω. Η άδεια πατρότητας, ε, η οποία ακούγεται τα τελευταία χρόνια, είναι για κάτι αρκετά καινοφανέ, το οποίο φαίνεται να αποκτά μεγάλη δημοτικότητα. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Από πλευρά ίσων δικαιωμάτων, εσείς ω εμπειρογνώμων, πώς βλέπετε το θέμα της άδεια πατρότητας. Για να είμαι πιο όμω, θεωρείτε ότι είναι ίση αξία ε, με την άδεια μητρότητας. Θα πρέπει να θεωρείτε ω υποκατάστατο κάτι που μπορεί να υποκαταστήσει την ε, άδεια μητρότητα ή θα μπορούσε να είναι ένα συμπληρωματικό στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να συμπληρώσει και να εμπλουτίσει την ίδια την άδεια μητρότητας. Η άδεια πατρότητας λοιπόν είναι γιατί πρέπει να καλύπτονται κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ίδια την άδεια μητρότητας. be... Νομίζω ότι στόχος μας θα πρέπει να είναι οι γονείς γονείς παιδιών που μπορεί να μην είναι πάντα ένα άνδρας και μια γυναίκα να μπορούν να μοιράζονται την άδεια του γονιού. Εγώ θα ήθελα να την ε, ε, αποκαλούμε έτσι, άδεια γονέα. Και αυτό θα πρέπει να είναι και ο στόχος μας. υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις στις οποίες ε, τα έσοδα των γυναικών είναι πολύ λιγότερα από των ανδρών και αν δεν αποζημιώνεται κάποιος ε, στο σύνολό του για τον χρόνο άδεια που παίρνει, τότε υπάρχει μεγάλη οικονομική απώλεια για οικογένειες τις οποίες οι γυναίκες δεν πληρώνονται το ίδιο με τους άνδρες. Όλα αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Αν δεν υπάρχει λοιπόν ίση μεταχείριση στους μισθού, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε και ε, ίσο καταμερισμό των γονικών αρμοδιοτήτων, αν θέλετε. Θα πρέπει όλα αυτά λοιπόν να συνεργάζονται και να μην τα επιβλέπουμε ως μεμονωμένα τμήματα. Ευχαριστούμε κυρία Κέλλη ε, για τις απαντήσεις. Η κυρία Κώστα θα, βάλει, θα θέσει την ε, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κέλλη για την παρουσίασή της. Να τη συγχαρώ και για το πάθος που τη διακρίνει για ένα θέμα που αφορά τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών. Θεωρώ και εγώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα Ινστιτούτο το οποίο θα έχει ένα συμβουλευτικό φόρουμ το οποίο θα μπορεί να εξετάζει όλο το φάσμα των θεμάτων που αφορούν στις γυναίκες και, και τους άνδρες φυσικά, γιατί νομίζω ότι η πιο σημαντική επισήμανση που κάνατε είναι ότι θα πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά και από την οπτική των ανδρών ε, και όχι μόνο για τις γυναίκες. Κατά την άποψή μου είναι μια, ένα από τα πρώτα θέματα που θα πρέπει να διαβιβάσει το Ινστιτούτο, ότι ασχολείται και με τα δύο φύλλα και με την προοπτική να καθορίσει ποια είναι τα χάσματα των δύο φύλων στα θέματα πολιτικής. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μου φαίνεται ότι ένα από τα σημεία στα οποία εστιάζει η δράση του φόρουμ ε, ως προς το συμβουλευτικό του ρόλο θα πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε, δεδομένου ότι μιλάμε και για 27 ε, χώρες, το θέμα της σύγκρισης των ε, στατιστικών που αφορούν στην ισότητα των φύλων, των ε, δραστηριοποιούμενων οργανισμών. Αυτή τη στιγμή στις διάφορες χώρες διαπιστώνουμε μία πτώση στην αποτελεσματικότητα και στο ρόλο αυτών των οργανισμών. Και θεωρώ ότι αυτοί οι οργανισμοί περιμένουν αυτό το Ινστιτούτο ως ε, μια τεχνική συνδρομή που θα τους βοηθήσει να εφαρμόσουν και να κάνουν και μια αντιπαρέθεση των πολιτικών. Χρειαζόμαστε δηλαδή όχι μόνο την εφαρμογή αλλά και την επαλήθευση του πώς ε, τα θέματα της ισότητας των φύλων εφαρμόζονται ε, στις χώρες μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια προοπτική πραγματικά μακρόπνοη ε, που θα έχει βέβαια και κάποιες εξειδικεύσεις σε κάποια σημεία. Δεν ξέρω αν συμμερίζεστε την απόψή μου, αλλά είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε ιδιαίτερως να επισημάνουμε. Ευχαριστώ να μας απαντήσει η Λίζ. Ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε κάποιους ε, βασικούς δείκτες. Αλλά πέρα από αυτούς, ε, η ίση μεταχείριση στους μισθούς, η ίση επασχόληση, η ίση συμμετοχή, χρειαζόμαστε και ένα ευρύτερο ε, σύνολο δικτών για τους οποίους θα πρέπει να μας δίνουν στοιχεία όλες οι χώρες. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση. Υπάρχουν ε, σχετικές αιτήσει και από το Ηνωμένα Έθνη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Συμβούλιο της Ευρώπης για στατιστικά στοιχεία τα οποία θα κάνουν καταμερισμό των φύλων εδώ και δεκαετίες και οι πολλές χώρες ε, μεταξύ των οποίων και η δική μου δεν τα δίνουν αυτά τα στοιχεία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ένα μέσο το οποίο δεν θα είναι ιδιαίτερα ε, Επαχθέ, αλλά ταυτόχρονα θα μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνουμε τα στοιχεία που θέλουμε και ε, θα μπορούμε να συγκρίνουμε και ίσως προς ίσω. Διότι πολλές φορές ο τρόπος με τον οποίο συντάσσονται τα στατιστικά στοιχεία ε, είναι τόσο διαφορετικά που ουσιαστικά δεν συγκρίνουμε τα ίδια πράγματα. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν μόνο δείκτε, χρειαζόμαστε και ε, ένα κοινό τρόπο καθορισμού ε, των διαφόρων στοιχείων και τα δεδομένα να δίνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα μαζί σα. Επίση θα πω ότι ένα από τα πράγματα που χρειαζόμαστε είναι και οι έννοιε οι οποίε θα μα βοηθήσουν να διαπιστώσουμε ότι δεν μιλάμε μόνο για άνδρες και γυναίκε. Θα πρέπει να μιλάμε για ε, καθεστώτα που φορούν στο φύλλο, ε, να μην υπάρχει δηλαδή ένας ανταγωνισμός και να λέμε ότι δεν μιλάμε αρκετά για τους άνδρες ή μιλάμε πολύ για τους άνδρες. Αυτό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι η αλληλοσύνδεση μεταξύ ανδρών και γυναικών και τι αποτελέσματα προκύπτουν σε θέματα ισότητας ή ανισότητας. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Να υπάρχει ένα λεξιλόγιο, μια ορολογία που θα μας επιτρέπει ε, να αποφεύγουμε τις περιττές συζητήσει για το τι είναι ή δεν είναι ε, το φύλλο και οι διαφορές του. Σας ευχαριστώ εκ μέρους ε, Επιτροπής μας, κυρία Κέλλη, για την παρουσίασή σας και για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Νικόλα Ταμπίτου, Νικολέτα Μπίτου, η οποία είναι η συντονίστρια του κέντρου ΡΟΜ στο Την καλωσορίζω θερμά στην Επιτροπή μας και ελπίζω ότι ε, ε, θα μας πείτε ποιες είναι οι εμπειρίες σας σχετικά με ε, την ισότητα των φύλων και πόσο θα μπορέσετε να συμβάλλετε στο φόρουμ εμπειρογνωμόνων. Θα κάνετε μία σύντομη παρουσίαση και μετά θα έχετε ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής. Καλησπέρα. Δεν χρειάζεται να ξαναπαρουσιαστώ εφόσον η κυρία Πρόεδρος ούτως ή άλλως το ε, έπραξε θα σας παρουσιάσω την εμπειρία μου στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών ε, διότι εδώ και 18 χρόνια είμαι δραστήρια στο συντονισμό των υποθέσεων των ΡΟΜ ε, τελείωσα τις σπουδέ μου το 1997 και εδώ και 10 χρόνια ασχολούμαι εντατικά με το να προωθώ την, ε, το πρόγραμμα των διεθνών οργανώσεων και όχι μόνο. Οπότε το 1999 άρχισα να καταρτίζω για το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, μία έκθεση για την κατάσταση των ΡΟΜ ε, στις χώρες ε, των κρατών μελών του Συμβουλίου και το εξετάστηκε στο Συμβούλιο Υπουργών και απετέλεσε την αρχή της δουλειάς μου, τη βάση της δουλειάς μου επί 10 χρόνια. Δηλαδή παρακολούθησα τις συστάσεις τις οποίες είχα περιλάβει στην έκθεσή μου για να υλοποιηθούν και αυτό πολύ πεισματικά. Παρακολούθησα λοιπόν το Συμβούλιο της ε, Ευρώπης, επίσης προσέφυγα στα Ηνωμένα Έθνη με διάφορους τρόπους για να μπορέσω να ε, προωθήσω τη θέση των γυναικών ε, στο Πεκίνο συν 5, Πεκίνο συν 10. Έχω ασχοληθεί με θέματα της ισότητας των φύλων στις διάφορες αυτές οργανώσεις και σε επίπεδο του ΟΗΕ συμμετέχω στους εμπειρογνώμονες για την ισότητα των φύλων για την προετοιμασία του συνεδρίου του Ντόρμπαν Είναι η πρώτη ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα ασχοληθεί ε, με την ε, ισότητα των φύλων και τις διακρίσεις στα επίπεδα του ΟΗΕ ε, άλλωστε έχω συνεργαστεί με τον ΟΑΣΕ ε, και ε, επίσης σε με έναν οργανισμό ο οποίος προωθεί τα θέματα των ΡΟΜ και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εκεί εξετάζουμε και τα συστατικά της ισότητας των φύλων. Ε, ε, ε, έχω συμμετάσχει και στον αγώνα για την καταπολέμηση του εμπορίου λευκής αρκός και Ε, τα, οι διάφοροι οργανισμοί που ασχολούνται με τους ε, ΡΟΜ έχουν προβεί σε έρευνες σχετικά με τη σωματεμπορία και έχουν ε, ξεκινήσει μία εκστρατεία κατά της σωματεμπορίας. Άλλωστε Έχω συμμετάσχει και στην ε, δεκαετία για την ε, ένταξη των ε, ΡΟΜ όπου πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή και προωθούν την ισότητα των φύλων. Γι' αυτό και έχει καταρτιστεί ένα πρόγραμμα δράσης για τη δεκαετία. Αλλά δυστυχώς η εφαρμογή του προγράμματος αυτού, ιδίω όσον αφορά την ισότητα των φύλων, δεν έχει προχωρήσει και τόσο πολύ. Δεν είχε τόση επιτυχία. Και βεβαίως πολύ σημαντικό είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχω προωθήσει εδώ και πολλά χρόνια την έκθεση για τους ΡΟΜ που υιοθετήθηκε το 2006. Είχα συμμετάσχει και στην ακρόαση που οργανώθηκε σχετικά με την έκθεση αυτή. Ε, έχω ασχοληθεί και με την έκθεση ε, για την απασχόληση των γυναικών εις ε, την ε, κεντρική και ανατολική Ευρώπη για να καλύπτω την πτυχή της χώρας μου και επίσης ε, προώθησα την έκθεση για την κατάσταση της απασχόλησης γυναικών ε, ΡΟΜ. Ε, πέραν αυτού έχουμε κινητοποιήσει διάφορες ε, γυναίκες ε, σε ε, ρουμανικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να μπορέσουν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους και συντονίζω και ένα άτυπο δίκτυο 15 χωρών όπου έχω κάνει πολλές έρευνες μέσω του δικτύου αυτού. Το δίκτυο λοιπόν αυτό που ανέφερα είναι πολύ δραστήριο ακόμη και αν είναι άτυπο. Πρόκειται για μια διεθνή οργάνωση. Είμαι επίσης μέλος του λόμπι των ε, ε, Ρουμάνων γυναικών και πέραν αυτών Ε, η κινητοποίηση των γυναικών ΡΟΜ είναι πολύ μεγάλη διότι θέλαμε να προωθήσουμε τα δικαιώματά μας πράγμα το οποίο δεν ήταν εύκολο και κάναμε έναν αγώνα για να πείσουμε τους άντρες μέλη ε, της Επιτροπής Ισότητας των φίλων ότι και οι γυναίκες ε, ε, δικαιούνται κάτι περισσότερο Επίσης όσον αφορά την κίνηση ΡΟΜ έχω συντονίσει διάφορες ομάδες με την ρουμάνικη πτέρυγα και αυτές είναι ουσιαστικά οι δραστηριότητές μου. Προσπάθησα να δημιουργήσω γέφυρες μεταξύ διαφόρων ομάδων και διαφόρων κινήσεων και στην αρχή δεν ήταν εύκολο να συμμετάσχει κανείς ε, εις ε, την κίνηση αυτή και να θέτει τα ερωτήματα που σχετίζονται με τις γυναίκες ΡΟΜ. Εις ε, το φόρουμ των εμπειρογνωμόνων πιστεύω ότι θα μπορέσω να συμβάλλω διότι εν ονόματι της ε, οικονομικής ε, κρίσης οι κυβερνήσεις μειώνουν τον προϋπολογισμό τους και ε, οι πρώτες οργανώσεις που πλήττονται είναι οι οργανώσεις ισότητας των φύλων. Παίρνω σαν παράδειγμα την Ρουμανία η οποία έκλεισε τον οργανισμό για ισότητα ανδρών και γυναικών και σκοπεύει να διαλύσει και την Επιτροπή του Κοινοβουλίου που ασχολείται με αυτό το θέμα. Σε τέτοιο λοιπόν πολιτικό περιβάλλον πιστεύω ότι πρώτες θα πληγούν οι γυναίκες και οι περιθωριοποιημένες ε, ε, ομάδες και γι' αυτό ήθελα να παρουσιάσω αυτό το θέμα και ε, να τους εξηγήσω ποια είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Δεν, υπάρχουν, μόνο, δεν υπάρχει μόνο ένα είδος ε, γυναικών ε, που ζουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη αλλά υπάρχει, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την Ισότητα των Φύλων το 2008 έδειξε ότι το κενό μειώθηκε από 17% στο 14%. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες ακόμη που δεν έχουν μία τακτική εργασία και προτείνω να συγκεντρωθούν στοιχεία τα οποία να βασίζονται στην ηλικία διότι τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουν ε, συγκεντρωθεί δεν είναι ε, ενοποιημένα όσον αφορά την ηλικία Ίσως λοιπόν ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα έπρεπε να συγκεντρώσει στοιχεία αυτού του είδους και να συγκρίνει γυναίκες διαφορετικών ομάδων, εθνικές μειονότητες, ανήπαντρες μητέρες, ε, μετανάστες ε, δευτέρας ή τρίτης γενιάς που αντιμετωπίζουν προβλήματα για πρόσβαση όχι μόνο στην ε, εργασία αλλά και στα, μέσα στην ε, κοινωνία τους όπου υπάρχουν περιορισμοί και βία που επηρεάζει τις γυναίκες αυτές και νομίζω ότι μπορώ να είμαι ο άνθρωπος που πάντοτε θα προωθεί τα θέματα αυτά διότι γνωρίζει ότι η ζωή των Ευρωπαίων πολιτών αυτή, αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο εύκολη. Θα σταματήσω εδώ, θέλω όμως να πω ότι ο ρόλος και η συνεργασία με τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ βασικός για να μπορεί κανείς όπως προβλέπεται από την εντολή να προωθήσει την κατάργηση των στερεοτύπων. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο να συμβάλλουμε στην προσπάθεια, αλλά να ασχοληθούμε και με τις ε, γυναίκες οι οποίες έχουν υπερβεί τα όρια της, τους, της κοινότητάς τους. Είναι πολύ δυσχερής η εργασία αυτή. Έχουμε εργαστεί πολύ ε, για τα μέρα της ενημέρωσης και η πείρα μου πιστεύω μπορεί να είναι χρήσιμη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπιτού πραγματικά για την παρουσίασή σας. Ε, τώρα θα ακούσουμε ε, τα μέλη της Επιτροπής. Η κυρία Γιαβόκα νομίζω ζήτησε πρώτη το λόγο για να θέσει ερωτήματα στην υποψήφια. Ευχαριστώ ε, κυρία Μπιτού για την παρουσίαση που κάνατε. Ανέκαθεν μας ε, βοηθούσατε εδώ στην Επιτροπή ε, Γυναικών για να κατανοήσουμε αυτά τα περίπλοκα προβλήματα. Κάτι που δεν είχαμε χρόνο να συζητήσουμε στην ακρόαση και στη, μέχρι να εκπονήσουμε την ίδια την έκθεση επειδή μιλάτε για τις γυναίκες ε, Ρώμα ως κομμάτι της κοινωνίας της Ρουμανίας αλλά ποτέ δεν συζητήσαμε ποιε είναι οι βασικές προκλήσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν ε, ε, γενικότερα γυναίκε που, ε, που ανήκουν σε μειοψηφίε, όπως οι γυναίκε ΡΟΜ. Δηλαδή, μπορείτε να μας πείτε περισσότερα πράγματα σχετικά με, την, με το πώς μπορούμε να προβάλλουμε αυτά τα ζητήματα, αποκτήσουμε μεγαλύτερη δημοσιότητα χάρη στο Ινστιτούτο. Ε, σας ευχαριστούμε κύριε Γιαβόκα. Κυρία Μπιτού, θα θέλατε να απαντήσετε. Είναι δύσκολο το ερώτημά σας. Ε, προσπαθώ να το απαντήσω εδώ και 10 χρόνια. Προσπαθώ δηλαδή να ε, βρω ε, την πλέον εξισορροπημένη διατύπωση για να το εκφράσω δημόσια, να εκφράσω δημόσια αυτή την άποψη στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν ισχύουν τα ίδια δεδομένα για όλες ε, τις κατηγορίες. Ε, Μέσα στην κοινότητα Ρώμη υπάρχουν πολλές υποκατηγορίες, για να το πω έτσι. Ε, οι γάμοι που γίνονται σε πολύ νεαρή ηλικία. Να ένα βασικό θέμα που καλείται να αντιμετωπίσει η κοινότητα Ρώμ και μόλις τώρα συνέταξα ε, την τελική έκθεση για αυτούς τους γάμους σε μικρή ηλικία στη κοινωνία των ε, ΡΟΜ που θα, και η έκθεση θα δημοσιευτεί μέσα στο επόμενο εξάμεινο. Τώρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Ε, ακραία ένδια άλλο πρόβλημα που πλήττει τις ε, κοινότητες αυτές ε, στην Ανατολική Ευρώπη υπάρχουν ε, αστικές κοινότητες καλά ενταγμένες στην κοινωνία που υφίστανται διακριτική μεταχείριση και ας το πούμε έτσι, και έχουν χάσει διάφορα στοιχεία της κουλτούρας τους, δεν μιλούν τη γλώσσα κτλ. έγιναν οι μαύροι της Ευρώπης. Ε, ας κάνουμε αυτή τη σύγκριση. Δεν έχουν διατηρήσει τις πολιτιστικές τους ε, συνήθειες, ε, τις παραδόσεις τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το πρόβλημα διότι όσοι ε, κάποιοι τους δίνουν δάνεια και στη συνέχεια αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν τα δάνεια εξαρτώνται από τους δανειοδότες. Υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα. Πώς ακριβώς τώρα να το ρυθμίσουμε το πρόβλημα. Κοιτάξτε, ε, πρέπει να εγγραφεί στο πρόγραμμα εργασιών, να συνειδητοποιήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που ε, αντιστοιχούν όλες, ε, που συγγνώμη, απασχολούν όλες τις μειοψηφίες και όχι την ε, πλειοψηφία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσχάτως στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, σκοτώθηκε μία νέα γυναίκα. ήταν ένα έγκλημα τιμής, τη σκότωσε ο πατέρας της. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την κοινότητα των Ρώμ, ισχύει και για κάποιες μουσουλμανικές κοινότητες. Εγώ δυσκολεύτηκα για να βρω τρόπο να μιλήσω δημόσια για αυτά τα ζητήματα σε επίπεδο εκπόνησης πολιτικής και σε επίπεδο ανάλυσης των εθνικών πολιτικών, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε κατά πόσο τα κράτη-μέλη ε, ασχολούνται με το ζήτημα της ισότητας των δύο φυλών, αλλά για όλες τις γυναικείες πληθυσμιακές ομάδες. Εάν αποδίδουμε σημασία σε κάποια ζητήματα, έμεσα πλήττονται ε, κάποιες ομάδες ε, που παραμελούμε όπως ε, η ΡΟΜ. Για το 2010 τώρα, έτος καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, το Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων οφείλει να διαδραματίσει σημαντικότατο ρόλο για να κάνει μια εκστρατεία ενημέρωσης όπου θα προβάλλονται οι μειοψηφίε ε, της κοινωνίας μας ε, και άλλες πληθυσμιακές ομάδες που αποκλείονται κοινωνικά. Αυτό νομίζω ε, θα έχει πάρα πολύ θετική επίπτωση σε αυτές τις κοινότητες. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Σαμπόφσκα τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Αμπιτού, σας θυμάμαι πολύ καλά. Έχετε επισκεφθεί και στο παρελθόν την Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι αυτά που μας είπατε εδώ σήμερα καταδεικνύουν ότι έχετε μία μακρόχρονη πείρα σε ένα από τα πιο δύσκολα θέματα τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων μας και είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει και με την κοινωνικό αποκλεισμό, την ένδια, την ε, δημόσια υγεία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά θέματα που σχετίζονται με αυτό το βασικό θέμα. Ε, τα ακούσαμε και στην παρουσίασή σας και θα ήθελα να κάνω την εξής ερώτηση. Ποια θεωρείτε ότι θα πρέπει να είναι τα καθήκοντα του Ινστιτούτου σε θέματα φύλου. Θα πρέπει απλά να συλλέγει πληροφορίες από τα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα αναλύει και κατόπιν να τα παρουσιάζει. Είτε αυτό είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι σε γραπτή μορφή μέσω εκθέσεων και να επαναλάβω εδώ ότι μας ενδιαφέρει και η προβολή του στα μέσα ή θεωρείτε ότι θα πρέπει να εστιάζει κυρίως σε κάποιες ε, ενεργές στρατηγικές πολιτικές σε θέματα ισότητας των φύλων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σαμπόσκα. Κύριε Μπιτού, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα, παρακαλούμε. Αν ήταν στο χέρι μου, θα ήταν και τα δύο. Εγώ θα ήθελα να επιλέξω και τα δύο. Αν δω το κατάλογο των καθηκόντων του Ινστιτούτου, Νομίζω ότι το Ινστιτούτο έχει να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο τόσο στη συλλογή των δεδομένων και την παρουσίασή τους ε, στο κοινό, αλλά θα πρέπει να συνεισφέρει και με άλλους δείκτες και μεθόδους συλλογής δεδομένων, όπως ε, για παράδειγμα κάνει Eurostat μέχρι τούδε. Χρειαζόμαστε λοιπόν άλλες μεθόδους και άλλους δείκτες για τη συλλογή δεδομένων ε, που θα βοηθήσουν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τα κράτη-μέλη να κατανοήσουν λίγο καλύτερα πώς έχει η, πραγματική, η πραγματικότητα. Διότι σε κάποιες περιπτώσεις διαβάζω οδηγίες, συστάσεις, εκθέσεις που μου δίνουν την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο κενό μεταξύ των ε, διατάξεων των εγγράφων αυτών και της ε, πραγματικότητας ε, που διαπιστώνω εγώ επιτόπου δυστυχώς καθημερινά. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για το Ινστιτούτο να συλλέγει ε, δεδομένα όχι μόνο όμως διαμέσου των θεσμικών οργάνων αλλά και άμεσα από ανεξάρτητους φορείς και όχι μόνο από εθνικούς φορείς. Όσον αφορά τώρα την χάραξη πολιτικής, νομίζω ότι και πάλι μπορεί να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, διότι ε, ε, γράφουμε και διαβάζουμε ότι θα πρέπει να αναλύει μεθόδους, μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές. Μεταξύ των καθηκάντων του Ινστιτούτου λοιπόν είναι και αυτό. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να αναλυθεί και ο τρόπος με τον οποίο επί παραδείγματι πώς εφαρμόστηκαν οι πολιτικές ισότητας των φύλων ε, στο δεύτερο και τρίτο κύμα ε, ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πώς έχουν προχωρήσει τα πράγματα, για παράδειγμα, στις χώρες που εντάχθηκαν το 2004. Εκεί υπήρχε μεγάλη πίεση να υιοθετηθούν πολιτικές κατά των διακρίσεων και δεν ήρθανε μόνο εντός ενό πολιτικού μοχλού, πρόκειται για ένα από τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται για την ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε αυτό, ε, δημιουργήθηκαν θεσμοί, ε, υπάρχουν πολιτικές κατά των διακρίσεων, υπάρχουν πολιτικές ε, για την ισότητα των φύλων, αλλά νομίζω ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου οι πολιτικές αυτές δεν φαίνεται να συνδέονται και με μια πολιτική βούληση. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα, διότι μακροπρόθεσμα οι πολιτικές αυτές μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές. Ευχαριστούμε ε, κυρία Μπιτού. Εξ ονόματος της Επιτροπής σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας και για τις αφείς απαντήσεις που δώσατε. Ε, σας ε, καλωσορίζουμε και πάλι όποτε θελήσετε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε. Det är er en eh, glädje för Χαίρομαι που σήμερα καλωσορίζουμε την κυρία Ζινέβρα Κόντιο Ντορίζιο. Ε, είναι διδάκτορ ιστορίας πολιτικής σκέψης στη, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης και διευθύντρια του Διεθνούς κέντρου μελετών για τις γυναίκες, για ε, θέματα κοινωνίας και ιστορίας και επίσης ε, είναι και πολιτική επιστήμονας. Ε, και ασχολείται όλος ιδιαίτερος με τα ζητήματα που αφορούν στις γυναίκες. Καλωσορίσατε, θα σας ακούσουμε για 10 λεπτά περίπου μας κάνετε μια παρουσία σχετικά με την εμπειρία που έχετε στον τομέα της ισότητας των δύο φίλων και να μας εξηγήσετε ε, σε τι θα μπορούσατε να συνεισφέρετε, τι θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στο Ινστιτούτο και στο Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων. Κατόπιν θα σας κάνουν ερωτήσεις τα μέλη της Επιτροπής, αλλά προς το παρόν ακούμε την ε, παρουσίασή σας. To speak in French, okay. Θα μιλήσω στα γαλλικά αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπως είπατε, διδάσκω ιστορία πολιτικής σκέψης. Όταν άρχισα τη σταδιοδρομία μου, είναι πολύ δύσκολο τώρα να σας εξηγήσω όλη την σταδιοδρομία μου στον τομέα της έρευνας σε δύο λεπτά, αλλά θέλω να αναφερθώ τουλάχιστον σε δύο-τρία σημεία που έχουν σημασία για να καταλάβετε τι θα μπορούσα να συνεισφέρω σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Εφόσον διδάσκω ε, ιστορία πολιτικής σκέψης, όταν άρχισα την έρευνα μου, ε, άρχισα να συνειδητοποιώ ότι στα ε, δεν υπήρχε καμία θέση για τις γυναίκες ε, στον τομέα των, ε, της ε, ιστορίας πολιτικής σκέψης και άρχισαν να μελετώ τους διάφορους συγγραφείς για να δω ακριβώς τι έχουν πει για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Έκανα λοιπόν διάφορες έρευνες που όμως ε, με έφεραν σε δύσκολη θέση σε σχέση με τον ακαδημαϊκό κόσμο γιατί σε ακαδημαϊκό επίπεδο δεν ε, ε, θεωρεί το δογματικό το να κάνει κανείς τέτοια έρευνα. Ήταν λίγο περιθωριοποιημένη η μέθοδος. Εγώ συνέχισα αναπτύσσοντας μία μέθοδο, δεν θα ήθελα να δώσω εκεί όλο το βάρος, απλά για να καταλάβετε ποια είναι η σταδιοδρομία μου. Ε, Συνέγραψα βιβλία ε, για τους ε, νομικούς του σύγχρονου κόσμου και είδα ότι οι νομική του 17ου και 18ου αιώνα είχαν προβάλει μια περίεργη προσέγγιση του φεμινισμού στον τομέα του δικαίου. Ε, και στον ε, κόσμο της ε, πολιτικής σκέψης δεν είχαν καμία θέση ισχυρίζονταν οι γυναίκες. Εγώ απέδειξα το αντίθετο. Υπήρχε γυναικεία πολιτική σκέψη και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στο επίπεδο του κράτους ο άντρας μπορούσε να κυκλοφορεί ενώ η γυναίκα ήταν περιορισμένη στην ιδιωτική σφαίρα, στο σπίτι. Άρχισα να κάνω αυτές τις έρευνες και διαπίστωσα ότι ε, υπήρχαν πολλές γυναίκες που είχαν βρει τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτές τις επικρίσεις σε σχέση με τον παραδοσιακό τους ρόλο. Έκανα και εγώ μια αντιπαραβολή ανάμεσα στη γυναικεία και την αντρική πολιτική σκέψη που είχαν ασχοληθεί με το θέμα της γυναίκας στην κοινωνία και την νομική διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών. Αυτό έκανα σε πανεπιστημιακό επίπεδο και μεταξύ άλλων ήθελα να διαδώσω τις γνώσεις, τις γνώσεις που απέκτησα για να μην μείνουν θαμμένες όπως στο παρελθόν γιατί ε, ε διάφορες γυναίκες είχαν μελετήσει το θέμα αλλά δεν είχαν φροντίσει να διαδοθούν οι πληροφορίες. Από το 85 και μετά διδάσκω εκτός από την ιστορία της πολιτικής σκέψης ε, διδάσκω και την ιστορία της θέσης ε, των γυναικών. που μπορεί κανείς να εξετάσει από διαφορετικές ε, σκοπιές. Ε, εγώ δεν έχω όνειρο, έχω έναν εφιάλτη μπροστά μου. Βλέπω μία ολόκληρη γενιά φοιτητών που βγαίνουν από το πανεπιστήμιο χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για την ιστορία των γυναικών. Ενώ πρέπει να είναι κοινό κληροδότημα όλων από των αντρών και των γυναικών. Αν ναι, δεν υπάρχουν αυτές οι γνώσεις, δύσκολα μπορούμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων. Ακριβώς επειδή απουσιάζουν, ε, δεν, ε, υπάρχει έλλειψη αυτών των ε, γνώσεων. Δεν μιλώ για φεμινισμό, δεν μιλώ για τις παραδοσιακές συζητήσεις, αν είναι είσαι οι γυναίκες με τους άντρες κτλ. Σας μιλώ για την ιστορία της δημοκρατίας και την πρόσβαση των γυναικών στα πολιτικά δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη. Αυτές οι γνώσεις δεν είναι κοινέ, ε. είναι, ε, ε, εξακολουθούν, να, αποτελούν περιουσία των ειδικών. Δηλαδή σαν να μην έπρεπε η κοινωνία να είναι κάτοχος αυτών των γνώσεων. Στην Ιταλία γιορτάζουμε τα 150 χρόνια της ενότητας του έθνους και στην επέτειο αυτή κανείς δεν θα θυμηθεί τις γυναίκες που συνεισέφεραν ε, στην οικοδόμηση του έθνους. Ε, εγώ μόλις εξέδωσα ε, μια ανθολογία που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η ανθολογία της ευρωπαϊκής χειραφέτησης. Ισχυρίζονται κάποιοι ότι είναι πολύ δύσκολο να συντάξει κανείς ευρωπαϊκό εγχειρίδιο ιστορίας και συγκεκριμένα η χειραφέτηση των γυναικών είναι ένα θέμα που εξετάζω από ευρωπαϊκή σκοπιάς. Πέραν αυτού, έχω συνεργαστεί σε μεγάλο βαθμό με διάφορα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Έκανα την πρώτη μελέτη που ζήτησε το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, το 84 ε, με μια ομάδα από τη Γαλλία, ε, την Ολλανδία και τη Φινλανδία και είναι μια μελέτη που χρησιμοποιείται ως αναφορά για την θέση των γυναικών στην πολιτική ζωή της Ευρώπης. Και τέλος, γιατί δεν προλαβαίνω έτσι να τα αναφέρω όλα τα συνέδρια, όλες τις δραστηριότητε που έχω κάνει μου υπήρξα και αντιπρόεδρος της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ομάδας ε, για την ε, ε, κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση στην Ευρώπη και δημοσιεύσαμε και μία μελέτη όπου κατάφερα να εγγραφεί η αξία της ισότητας και να αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκή αξία πέρα από τη ε, δήλωση του 1789, τη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ε, υπάρχει και αυτή η αναφορά γιατί δεν ωφελεί ε, να έχουμε ένα μοντέλο κοινωνίας όπου έχουν πρόσβαση σε όλες τις επιστήμες, σε όλες τις ε, δουλειές στην πολιτική οι γυναίκες Ε, χωρίς να αναγνωρίζεται ε, η ισότητα των γυναικών. Μπορώ να σας τα δείξω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στα πανεπιστήμια να υπάρχει και πολιτική για την έρευνα που να ε, ε, ασχολείται με τις γυναίκες. Εάν δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα για τις γυναίκες, όπως και σε άλλους τομείς, είναι αδύνατο να προχωρήσουμε. Εγώ είδα τι υπάρχει από πλευράς ιστορικής τεκμηρίωσης. Γράφουν όλοι για το Μακιαβέλη. Μα εδώ και αιώνε μιλάμε για αυτόν, όλα τα ξέρουμε για αυτόν. Συνεχίζουμε όμως με τα συγγράμματα, επανερμηνεύουν τα γεγονότα, αλλά για την ιστορία των γυναικών πρέπει να ξεθάψω τα στοιχεία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρω εγχειρίδια για ε, τα ιστορικά στοιχεία, εγκυκλοπαιδικά λεξικά δεν υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επιστημονική έρευνα ένα κομμάτι των κονδυλίων να πηγαίνουν στην έρευνα των ζητημάτων που σχετίζονται με τις γυναίκες. Ε, είναι ένα κενό αυτό και πρέπει να καλυφθεί. Αυτά ε, έχω κάνει. Τώρα τι μπορώ να κάνω στο μέλλον για το Ινστιτούτο. Κοιτάξτε, ε, όταν άρχισα να βλέπω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία η Ευρώπη άρχισε να έχει μία πολιτική για την ισότητα των δύο φύλων, μου φάνηκε ότι ονειρευόμουν. Ε, γιατί έτσι νομιμοποιούνται τέτοιου είδου μελέτες που σας περιέγραφα και είναι με πολύ σημαντική σύνδρομη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπόν. Εγώ συνέχισα να ερευνώ και να μελετώ γιατί ε, ε, είμαι υπεύθυνη και για το διδακτορικό το μοναδικό στην Ευρώπη νομίζω σχετικά με τις γυναίκες και την πολιτική ως προς την ισότητα των δύο φίλων. Παρακολουθώ εκ του σύνεγγυ το θέμα αλλά γνωρίζω και τις δυσκολίες που υπάρχουν για να εκπονηθεί πολιτική ειδική για τις γυναίκες. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα κάνω θαύματα αλλά μπορώ να συνεργαστώ με το Ινστιτούτο στο πεδίο της, ε, του πολιτισμού, ε, ε, της επικοινωνιακής πολιτικής, της ισότητας των δύο φύλων, γιατί εστερνίζομαι αυτές τις αρχές και βρίσκω ότι από αυτά τα προγράμματα υπάρχει αυτή η έλλειψη, δηλαδή η συγκεκριμένη σχέση με τα θεσμικά όργανα, εάν δεν πάρουμε κάποια αντικειμενικά δεδομένα, έτσι, δεν σας μιλώ εδώ για ιδεολογικού χαρακτήρα συζήτηση, για πολιτικές συζητήσεις, σας μιλώ για δεδομένα. Ε, σαν να μελετούσαμε την ε, ε, ιστορία της Ευρώπης χωρίς να ξέρουμε πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Ε, στην ε, Ιταλία δεν ξέρουμε πότε άρχισαν να πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο, να φοιτούν στο πανεπιστήμιο οι γυναίκες, πότε πήραν την άδεια ε, να ασκούν, ε, να είναι ελεύθεροι επαγγελματίε, πότε άρχισαν να ασχολούνται με τις επίστημες, πότε καταργήθηκε η απαγόρευση που υπήρχε για την εξέβρεση του πατρός. Υπήρχε αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. για την ιστορία της ισότητας των δύο φίλων είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή καταργείται η απαγόρευση της αναζήτησης του πατρός. Καταλαβαίνετε πρόκειται για σεξουαλική ανοσία που προσφερόταν στους άντρες ε, και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να ερευνήσουμε. Δεν μιλάμε μόνο για την ημερομηνία ε, πρόσβαση των γυναικών ε, στα πολιτικά δικαιώματα. Μιλάμε για την ιστορία ολόκληρη τη δημοκρατίας ε, που πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τα δύο μισά του πληθυσμού, και τις γυναίκες και τους άντρες. νομίζω ότι τα ξεπέρασα τα 10 λεπτά. Υπάρχουν ερωτήσεις που μπορούν να σας απαντήσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Παλανόβα, ήθελα να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο για μία έκθεση σίγουρα ε, μάλλον για τη μελέτη για την οποία μας μιλήσατε σίγουρα, ε, όχι μόνο εγώ αλλά και πολλά άλλα μέλη της Επιτροπής μας θα ήθελα να τη δουν αυτή τη μελέτη στην οποία αναφερθήκατε. Η κυρία Παβανόβα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ένα λεπτάκι μόνο να είμαστε σίγουροι, έτσι για να βρούμε το σωστό κανάλι, να σας ακούει η κυρία Ντορίζιο. Εντάξει τώρα. Ευχαριστώ. Αυτά που είπατε ήταν πολύ ενδιαφέροντα και ιδίως με εντυπωσίασε ιστορική, το πολιτικό ιστορικό υπόβαθρο της δημοκρατίας και της ισότητας των φύλων. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, διότι το περασμένο Σάββατο έγινε ε, μια, ένα μεγάλο συνέδριο για ισότητα των φύλων στη Ρώμη ε, όπου εκπροσωπήθηκαν γυναίκες από 40 εθνικές ομάδες ε, μέσω των οργανώσεών τους. Ε, μπορείτε ε, να, να μας πείτε ε, τι έγινε εκεί γιατί του χρόνου προβλέπετε ότι θα κάνουν μία λευκή βίβλο και θα ήθελα να μας πείτε τι έχει γίνει για να μας πείτε πώς αυτό το θέμα μπορεί να προχωρήσει.

με συγχωρείτε. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Προφανώς μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και ε, αυτή είναι η ιδέα μου. Δεν πρέπει δηλαδή να περιοριστούμε μόνο σε τομείς οι οποίοι είναι κεντρικοί. Η ιδέα μου είναι ότι η πολιτική των, ε, της ισότητας των φύλων είναι περίπλοκη και αναφέρεται σε όλους τους τομείς. Οικονομικό, ο κοινωνικό και αυτό που μέχρι στιγμής μας έλειψε ήταν ε, η η μεταβίβαση διότι δεν είναι ένα θέμα το οποίο αναφέρεται μόνο στις γυναίκες αλλά στη δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ε, μία, μία βάση στην οποία, την οποία να συμμερίζονται όλοι. Σας ευχαριστούμε. Η κυρία Κώστα τώρα. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου την ε, καθηγήτρια Κόντι Οντορίζιο. Είναι πάρα πολύ γνωστή στην ε, Ιταλία, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης, ε, στο Ρώμη 3 και για τις σπουδές της. Είναι τιμή λοιπόν για μένα να σας γνωρίζω και σας χαιρετώ λοιπόν δημοσίως. Και από τα όσα μας είπατε καταλαβαίνουμε πόσο εις βάθος έχετε κάνει ιστορική έρευνα και για τα θέματα της συμμετοχής ε, των γυναικών στη δημοκρατία και ε, τους οργανισμούς στους οποίους συμμετέχετε για την προαγωγή των ίσων ε, ευκαιριών. Θα ήθελα λοιπόν επί τη βάση αυτής της πείρας ε, να σας ρωτήσω το εξής. Μιλήσατε για κάτι συγκεκριμένο στην ομιλία σας. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να συσχετίζεται και θα πρέπει να είναι και στόχος αυτός του ινστιτούτου και εδώ μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πρέπει να εκπροσωπούν το Κοινοβούλιο και τις σχέσεις του λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και με άλλους οργανισμούς και άλλα θεσμικά όργανα των διαφόρων κρατών μελών σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεισφέρετε από αυτή την έννοια, δεδομένης και της απόλυτης καινοτομίας αυτού του Ινστιτούτου και της ε, υποχρέωσης να εργαστεί για να εφαρμόσει συγκεκριμένες πολιτικές ε, που αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κυρία Κώστα και εσείς ε, είστε πολύ αφοσιωμένοι ε, στον τομέα αυτό. Είστε αγαπητοί μου φίλοι, σας γνωρίζω εδώ και πολλά ε, χρόνια και ευτυχώς μου θυμήσατε κάτι που παρέλειψα στην παρουσίασή μου. Δηλαδή, σε σχέση με τις προσδοκίες για το Ινστιτούτο, δεν περιμένει κανείς να επανεφεύγουμε τον τροχό. Ε, απλά ε, θα πρέπει να υπάρχουν σχέσεις με αυτά που γίνονται στην Ευρώπη. Παραδείγματο χάρη εγώ έχω συμμετάσχει ήδη σε δύο ε, ευρωπαϊκές διασκέψεις για την ισότητα των δύο φύλων με πανεπιστημιακούς από όλες τις χώρες που οργάνωσε το ring του Παρισιού ε, και ε, έχει αρχίσει να αναδεικνύεται σε μια ε, πανεπιστημιακή νομοσπονδία που μελετά το ζήτημα αυτό. Δεν μιλούμε για θεωρητικές συζητήσεις. Ο στόχος είναι εκπόνηση πολιτικής για κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, ούτω ώστε οι έρευνες που έχουν γίνει πριν από 30 χρόνια, χτες, σήμερα, αύριο, να ομαδοποιηθούν με την στήριξη του Ινστιτούτου ε, και τη Ομοσπονδία και για το ίδιο το Ινστιτούτο αποτελεί έρισμα η δουλειά και το δίκτυο που έχουν φτιάξει τα πανεπιστήμια ούτω ώστε να δούμε πώς σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα ανάλογα με τις ε, ε, ακαδημαϊκές δομές είναι δυνατόν να ε, επιφέρουμε καινοτόμα στοιχεία ε, στην έρευνα διδακτικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο ε, απο, να ε, ε, αποφυτεί κανείς από την, από νομική παραδείγματος χάρη χωρίς να γνωρίζει κανείς τίποτα για την ιστορία των γυναικών ή από τη φιλοσοφική. Πώς δηλαδή οι αστυνόμοι, οι δικαστές, οι εισαγγελείς θα εφαρμόσουν τους, τους νέους νόμους για τις γυναίκες αν αγνοούν παντελώς Ακόμη και το κριτήριο της ισότητας ε, των ε, ευχαιριών ε, είναι μια έννοια που αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει μόνο αν γνωρίζει τη δυσμενή μεταχείριση που είχαν υποστεί οι γυναίκες. Πρέπει να γνωρίζετε την, την ιστορία της πολιτικής για την ισότητα των δύο φύλων. Επίση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προβληθεί η ανάγκη να γίνονται απολογισμοί ε, σε σχέση με τι ε, δύο. ισολογισμοί μάλλον ε, για τα δύο φύλλα. Πώ θα το κάνουν αυτό οι οικονομολόγοι, αν μέσα στη νομική, στην ιατρική, στη σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο δεν διδάσκεται κάτι τέτοιο και στο δικό μου το πανεπιστήμιο. Γιατί είναι γνωστό το δικό μου πανεπιστήμιο, διότι υπάρχει ευαισθητοποίηση για αυτή την έλλειψη, αλλά ξέρετε, ένα, δύο μαθήματα υπάρχουν μόνο για τις γυναίκες. Οι γυναίκες και ο κινηματογράφος, καλό είναι αλλά δεν φτάνει και το δικό μου το μάθημα ε, που είναι στις πολιτικές επιστήμες. Οι... Σας λέω, όσοι σπουδάζουν νομικά, όσοι σπουδάζουν οικονομία, δεν έχουν ιδέα, αποφυτούν χωρίς να γνωρίζουν τίποτα. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ζητώ συγγνώμη ε, σε θέση να αποτροπιάζομαι με αυτά που συμβαίνουν. Πρόεδρος, καταλαβαίνουμε και εμείς έχουμε αντίστοιχη δέσμευση, ξέρετε όλες εδώ, ε, όλοι εδώ στην Επιτροπή Γυναικών. Ε, θέλω και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας γιατί βλέπω πόσο σημαντική είναι η έρευνα για να προβάλλεται η εικόνα των γυναικών και η ιστορία τους. Και συμφωνώ με αυτό που είπατε και εγώ είμαι πεπισμένη ότι θα, για να σημειωθεί πρόοδος ε, πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να κοιτάζουμε πίσω μας, ε, να ε, μελετούμε την ιστορία. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Απλά ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Αφενός πρέπει να αυξηθούν ε, οι επιστημονικές έρευνες για αυτό το θέμα και πρέπει να προβάλλουμε το ρόλο και την εικόνα των γυναικών στην ιστορία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ωραία. Το δεύτερο κομμάτι είναι πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα των ερευνών, ούτως ώστε να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. Ε, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μας απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ε, διότι όντως πρέπει κανείς ε, να δώσει να καταλάβετε ε, ότι όσοι ασχολούνται με την πρόθεση της δημοκρατίας πρέπει να καταλάβουν και την πρόθεση των δικαιωμάτων των γυναικών. Γι' αυτό και χρειάζεται πολιτική θέληση για την επιστημονική έρευνα. Έχω ένα διδακτορικό ερευνητικό και έχω και μία μαθήτρια η οποία κάνει ένα διδακτορικό. Άρα το Πανεπιστήμιο επενδύει σε αυτή. Δεν ξέρουμε όμως τι θα γίνει μετά, διότι η έρευνα αυτή δεν είναι αναγνωρισμένη, τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιό μου. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνέχεια πρέπει να μάχομαι ενάντια στα πικρά λόγια και τα αστεία των συναδέλφων που με θεωρούν πολύ θεωρητική και προσπαθώ να παραμείνω στον τομέα μου, στον τομέα της επιστήμης δηλαδή. Προτείνω λοιπόν και θα ήθελα να σας το δείξω, να σας δείξω την ανθολογία μου η οποία μόλις ε, η οποία μόλις ε, εξεδόθη ε, λέγεται περφύλο επερσένιο», δηλαδή σιγά σιγά βαθμιαία. Πρέπει λοιπόν να προτείνουμε ε, βήμα προς βήμα πρότυπα γυναικεία διότι τα κοριτσάκια κοιτούν την τηλεόραση και βλέπουν μόνο αυτές τις πολύ ωραίες ε, γυναίκες με βαθύ ντεκολτέ στις 4 απόγευμα που κάνουν περίεργα πράγματα και αυτή δεν είναι η αξιοπρέπεια της γυναίκας πρέπει να παρουσιάζεται ένα θετικός ρόλος και οι γυναίκες οι οποίες έχουν ε, πολεμήσει για τη χειραφέτηση του, του γένους τους ε, και του φίλου τους ε, όντως ήταν σημαντικές. Θα ήθελα να παρακαλέσω την Ελίζα αν είναι εδώ να πάρει το βιβλίο μου για να σας το δείξω μετά. Αυτό μπορεί να είναι ένα ευρωπαϊκό εγχειρίδιο, ένα πρότυπο για τις γυναίκες και τους άντρες της Ευρώπης γιατί ο φεμινισμός δεν είναι μόνο μια ιστορία για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες που υπεραμείνθηκαν αυτών των ιδεωδών και ε, εγώ που είμαι ιστορικός έδειξα ότι η κατάσταση αυτή υπήρχε πάντοτε. Υπήρξαν Γαλλίδες, Αγγλίδες, Ιταλίδες και ε, Αμερικανίδες με πολύ στενούς δελσμούς ακόμη και πριν από το διαδίκτυο. Ε, δεν ξέρω πώς επικοινωνούσαν αλλά είχαν πολύ στενές σχέσεις. Σας ευχαριστώ θερμά εξ ονόματος ε, της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίασή σας και καλή επιτυχία με ό,τι κάνετε στο μέλλον. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία και σε εσάς. Ehm, Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γκρένερ. Ε, ένα μέρος των συναδέλφων όπως και εγώ έχουμε ήδη συνεργαστεί με την κυρία Γκρένερ στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ξαναβλέπουμε, Λίζη. Ε, ήσασταν μέχρι τον Ιούλιο του 2009 συντονίστρια στην Επιτροπή μας, αντιπρόεδρος στη Διεθνή Σοσιαλιστική επί σειρά ετών. Έχετε ασχοληθεί με διάφορες εκστρατείες ε, για να σταματήσει η βία, παραδείγματο χάρη κατά των γυναικών. Ε, δραστηριοποιηθήκατε επίσης πάρα πολύ ε, για την μηδενική ανοχή για τη βία κατά των γυναικών και έχετε αναλάβει διάφορες πρωτοβουλίες στη Γερμανία για να, ξεκινήσουν, να ξεκινήσει η εκστρατεία της κόκκινης κάρτας για την πορνεία των κοριτσιών την παιδική πορνεία. Τέλος πάντων ε, η Λίζη Γκρένερ έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες και δράσεις. Ε, θα σου δώσω 10 λεπτά για την παρουσίασή σου. Ε, μίλησε μας για την εμπειρία σου και πες μας τι μπορείς να προσφέρεις στο Ινστιτούτο και στο Φόρουμ των Εμπειρογνωμών και γενικότερα στον τομέα και μετά θα ακούσεις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σήμερα βρίσκουμε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών. Πολλές φορές χρειάζεται κανείς να αποστασιοποιηθεί για να επιτύχει την ε, ισοτιμία και χαίρομαι που είναι εδώ η κυρία Ζαμπόρσκα διότι έχουμε πολλές κοινέ εμπειρίες αλλά βλέπω και νέα μέλη που θα προσφέρουν ε, νέες εμπειρίες. Γιατί έχω ε, θέση υποψηφιότητα για τη θέση αυτή εμπειρογνώμωνα εμπειρογνώμονα είναι διότι θεωρώ ότι είναι πολύ βασικό αυτό το νέο Ινστιτούτο να μπορέσει ε, να συγκεντρώσει τις εμπειρίες που έχουμε από εμπειρογνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμβάλλει σε μία γρήγορη ε, εξέλιξη του θέματος. Έχουμε εμπειρία εδώ και 15 χρόνια στην Επιτροπή από του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργήθηκε η ιδέα αυτή και εσείς στην Επιτροπή αυτή έχετε κάθε συμφέρον να καταλήξει σε μία αίσια εξέλιξη αυτό το Ινστιτούτο τότε είχαμε, ε, ε, ε, τότε είχαμε επιλέξει την πρόεδρο η οποία μπορεί να διευθύνει σωστά το Ινστιτούτο και πέραν ε, του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει και το Κοινοβούλιο να στηρίξει την δουλειά της διότι και η πρώτη της ε, έκθεση είχε ε, πολύ καλά αποτελέσματα. Πρέπει να σας πω ότι καταρχήν εγώ θα ήθελα οι πολλές διαπιστώσεις τις οποίες ε, έχουμε να μπορέσουν να εφαρμοστούν. Το η εφαρμογή, implementation είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Οι καλές προτάσεις θα πρέπει να επηρεάσουν τη ζωή των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, γι' αυτό θα κάνω ό,τι μπορώ για να ε, γίνει επιτυχές αυτό το Ινστιτούτο. Επίσης ε, είχα συνεργαστεί με, το μεγάλο συνασπισμό για να προχωρήσει αυτό το Ινστιτούτο και δεν θέλω εδώ να απαριθμίσω όλες τις εμπειρίες τις οποίες έχω συλλέξει σαν συνεισηγήτρια στο θέμα αυτό αλλά όπως σας είπα αυτό που είναι πολύ βασικό είναι οι εμπειρίες αυτές τις οποίες έχουμε να μπορέσουμε να τις προωθήσουμε διότι βλέπω ε, στο, ε, προς τα πίσω ότι με τη διεύρυνση το 2004 σαν Επιτροπή Γυναικών καταφέραμε ε, να υπάρχει άξια εκπροσώπηση γυναικών από τις νέες χώρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ευρεθούν σε ηγετικές θέσεις και πολιτικές αλλά και οικονομικές τις στηρίζουμε και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να διατυπώσουμε μία νέα συντονισμένη στρατηγική και ελπίζω ότι το Ινστιτούτο Ισότητος των Φύλων θα μπορέσει να διατυπώσει προτάσεις οι οποίες πολιτικά θα μπορέσουν να υποστηριχθούν για να εφαρμοστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο μέλλον λοιπόν θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα αυτό αλλά επιπλέον και το γεγονός ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα πρόβλημα το οποίο συνεχίζεται με διάφορες μορφές στις διάφορες χώρες στο παρελθόν είχαμε ε, καταφέρει να καταρτήσουμε το πρόγραμμα Δάφνη που ήταν ένα καλό όπλο και ελπίζω ότι με την Επιτροπή ε, εδώ θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την την καλή δουλειά που έχουμε κάνει ε, διότι συνενώσαμε όλες τις δυνάμεις, τις μη κυβερνητικέ ε, ε, επιτροπές και οργανώσεις και το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε ότι με τις κοινέ μας δυνάμεις θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να βοηθούμε τις γυναίκες στον αγώνα αυτό διότι διαπιστώνουμε ότι στο διαδίκτυο αναπτύσσεται και βία κατά των γυναικών ε, και παιδική πορνογραφία και θα πρέπει να ε, αντλήσουμε από τις γνώσεις του Ινστιτούτου και να διατυπώσουμε νέες προτάσεις. Ένας άλλος τομέας στον οποίο ε, πλέον πρέπει να έχουμε αποτελέσματα είναι στο θέμα της ίσης αμοιβή για ίση εργασία. Και εδώ έχει γίνει καλή προκαταρτική εργασία, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, υπάρχουν υπάρχουν εφαρμογές διαφόρων προγραμμάτων στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συγκροτήσουν ένα σύνολο στο Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και να αποτελέσουν ένα πρότυπο για τα κράτη-μέλη το οποίο θα μπορέσει να χρησιμεύσει και για την νομοθεσία στο να υπάρχει μία ενιαία βάση ε, και αυτό είναι ένα από τα καθήκοντα τα οποία θα πρέπει να προωθήσει το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων. Επίσης επειδή έχω μεγάλη εμπειρία και στο Κοινοβούλιο αλλά και σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις, εδώ δεν αναφέρομαι στις μη κυβερνητικές οργανώσεις μόνο. Έχω προωθήσει τα θέματα αυτά και στο Ευρωπαϊκό Λόμπι των Γυναικών και εις διάφορες οργανώσεις των Ηνωμένων Εθνών ή με πολλές επαφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα μπορούσε να είναι χρήσιμες ε, διότι πρέπει κανείς να ξέρει πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας χώρος πολύ γνώριμος και αυτό θα μπορέσει να βοηθήσει και το Ινστιτούτο Ισότητας των φίλων να έχει μια τέτοια γενική εικόνα και να μπορέσει να αναπτύξει αυτές τις εμπειρίες. Η τελευταία μου εμπειρία ε, επίσης δεν είναι αμεληταία διότι πριν δύο χρόνια ε, κατήρτισα μία, ε, μία επιχείρηση με έξι θέσεις θέσεις εργασίας για γυναίκες ε, και προσπαθώ από την άλλη πλευρά πλέον όχι πολιτικά αλλά πρακτικά να, να υλοποιήσω την βελτίωση των συνθήκων διαβιώσεως των γυναικών αυτών για να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και ε, να ε, συμβάλλουν στους στόχους του Ινστιτούτου. Ε, θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι γίνεται με ένα διεθνές συνέδριο γυναικών. Ήδη στο Πεκίνο ή στο συνέδριο είχαμε καταρτήσει σαφείς στόχους και ακόμη και αν έχουν περάσει 20 χρόνια αν ε, ε, κοιτάξω τώρα μπροστά ως το 2015 πιστεύω ότι θα πρέπει το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων να συμβάλλει στην υλοποίηση ε, μίας ενός Ευρωπαϊκού Συνεδρίου ή ένα παγκόσμιο συνεδρίου για την ισότητα των φύλων. Πιστεύω ότι υπάρχει στήριξη για αυτά τα θέματα και το γενικό ερώτημα αν μπορεί ο κόσμος να επιλύσει την οικονομική κρίση και με υποπίες προϋποθέσεις θα επιτρέψει να αξιολογήσουμε ε, τα ε, διάφορα θέματα διότι οι γυναίκες ε, πρέπει να αναλάβουν το φορτίο της καθημερινής εργασίας ή αν χαθεί ένας πόλεμος οι γυναίκες είναι οι πρώτες που υποφέρουν τέλος πάντων υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν και να προωθηθούν πιστεύουμε ότι και σε εθνικό και σε διεθνές ε, επίπεδο, πανεπιστημιακό ή κοινωνικό έχουμε καλά αποτελέσματα στα οποία να βασιστούμε και το Ινστιτούτο το οποίο θα έχει περιορισμένο προϋπολογισμό εάν κοιτάξουμε τώρα τα ποσά που θα διατεθούν στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης θα χρειαστεί μία μικρή ομάδα, ένα μικρό διοικητικό συμβούλιο και μια ομάδα εμπειρογνώμων που θα εργάζονται ανεξάρτητα αλλά θα πρέπει να επιτύχουν σαφείς στόχους. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα των εμπειρογνωμόνων με την εμπειρία την οποία ε, έχω συγκεντρώσει διαμέσου των ετών και νομίζω ότι ε, με την ε, πολιτική μου εμπειρία θα μπορέσω να συμβάλλω στην επιτυχία επιτυχία του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φίλων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος θέλει το λόγο, παρακαλώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες θα κάνει την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να καλωσορίσω τη Λίζη σε αυτή την επιτροπή που ούτως ή άλλως είναι και δικό της κομμάτι, δικό της παιδί διότι δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι το πέρασμά της από την Επιτροπή ε, μας επέτρεψε να διεξάγουμε πολλές από τις εργασίες που μπορούν να κάνουν οι Ευρωπαίες γυναίκες ε, σε θέματα ισότητας σε κάποιες βαθμές είναι ένα συν το να γνωρίζει κανείς ε, το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να γνωρίζει τα θεσμικά όργανα, τους μηχανισμούς εργασίας και τι κανόνες μπορούμε να θεσπίσουμε για συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, αυτού του Οργανισμού Ισότητας που θεωρώ ότι είναι θεμελιώδης. Υπάρχουν θέματα τα οποία ανέφερε, τα οποία θεωρούμε ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά, όπως είναι η καταπολέμηση της βίας, ε, ε, κανόνες ισότητες προκειμένου οι γυναίκες να μπορέσουν να ενταχθούν όχι μόνο στην πολιτικό βίο αλλά και στην κοινωνική ζωή, στην οικονομική ζωή είναι θέματα τα οποία εξελίσσονται από τα διάφορα Ινστιτούτα, τους διάφορους οργανισμούς και ε, τα όσα θα μπορέσει να κάνει το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων είναι ε, πολύ σημαντικά, κυρίως ως προς την όθηση που μπορεί να δώσει. Θα ήθελα να ξέρω τι πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων όχι μόνο προς την αναζήτηση ισορροπία συμμετοχής μεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και για να μπορέσουμε να ε, πάυσει να υπάρχει αυτή η κρυστάλλινη οροφή. Ε, όταν λοιπόν οι γυναίκες αρχίζουν να συμμετέχουν στον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό βίο, αλλά δεν καταφέρνουν να φτάσουν στα ίδια επίπεδα εκπροσώπησης. Ε, ένα σαφές παράδειγμα το έχουμε εδώ, στο Κοινοβούλιο από την αρχή της κοινοβουλευτικής ζωής ε, άρχισε σιγά σιγά να αυξάνεται η συμμετοχή των γυναικών αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μια κρυστάλλινη οροφή που προϋποθέτει ότι την ε, πλειοψηφία των, ε, της Προεδρίας και της Αντιπροεδρίας των Επιτροπών της έχουν άνδρες κατά βάση ε, τις αντιπροσωπείες έχουν άνδρες κατά βάση τα ίδια τα θεσμικά όργανα δεν έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να προβλέψουν τη συμμετοχή των, των γυναικών. Και όπως και στην ε, πολιτική το ίδιο συμβαίνει και με τα συνδικάτα και τις επιχειρήσεις. Είναι αλήθεια, οι γυναίκες ε, ενσωματώνονται αλλά πρέπει ακόμα να σπάσει αυτός ο κρυστάλλινος ε, θόλος και να μπορέσουμε να συμμετέχουμε περισσότερο στα θέματα αυτά. Επίσης υπάρχει και ένα πολύ θεμελιώδες ζήτημα όταν συζητάμε για θέματα βίας γυναικών, για θέματα διαφοράς μισθών μεταξύ ανδρών και γυναικών, όταν συζητάμε όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ομογενή και κοινά κριτήρια τα οποία θα μας επιτρέψουν να κάνουμε μια πραγματική σύγκριση ως προς την ομοθεσία μεταξύ χωρών και ούτε καθεξής. Όταν μιλάμε για βία σε θέματα φύλου, κάθε χώρα χώρα έχει καθορίσει διαφορετικά κριτήρια. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να γίνουν οι συγκρίσεις. Είναι πολύ δύσκολο να εξετάσουμε και να γνωρίζουμε κατά πόσον η νομοθεσία που εφαρμόζει μια χώρα ε, ευνοεί την αλλαγή της πραγματικότητας. Ένας λοιπόν από τους βασικούς ρόλους που θα πρέπει να έχει το Ίδρυμα, ε, το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων είναι ε, να έχουμε ομογενή κριτήρια, ώστε όταν μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα να μπορούμε να έχουμε μια πολύ σαφή και πραγματική εικόνα ε, του πώς έχει η κατάσταση. Όπως σας λέω δεν είναι μόνο θέματα της καταπολέμησης της βίας ε, κατά των γυναικών ε, αλλά μπορεί να είναι και η διαφορά των μισθών ή οποιοδήποτε θέμα το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει μια πολιτική ισότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στη Λίζη για να μας απαντήσει. Ευχαριστώ. Μπορώ απλούστατα να συμφωνήσω. Χρειάζομαι κοινού δείκτες τους οποίους να μπορούμε να διαβάσουμε για να να δούμε πώς έχει εξελιχθεί η ισότητα διότι υπάρχουν ενάψματα και αυτό ακριβώς ε, περιμένω από το Ινστιτούτο ισότητα των Φύλων να ακολουθήσει αυτή την πορεία και ε, να ε, συνεργαστεί με τα Εθνικά Ινστιτούτα για να έχουμε κοινούς δείκτες και να μπορέσουμε να αποδείξουμε ότι δεν είναι μόνο ένα θέμα που απασχολεί στις γυναίκες αλλά είναι ένα θέμα στο οποίο θα, το οποίο θα υιοθετήσουν και οι άνδρες ε, υπεύθυνοι λήψεως αποφάσεων και ε, αυτό απεδείχθη ε, κατά την τελευταία επίσκεψή μας στη Σουηδία. Δηλαδή υπάρχει ένα συλλογικό, μια συλλογική συνειδητοποίηση η οποία αλλάζει στη Σουηδία ένας πατέρας ο οποίος οποίος ε, ε, δεν ε, δεν ασχολείται με την οικογένειά του και τα παιδιά του αρχίζει να προκαλεί την αποτροπή των συναδέλφων του και στη ε, Ισπανία υπάρχει αυτή η πολιτική ε, πρόοδος. Ε, μπορέσαμε να προωθήσουμε την νομοθεσία. Έχουμε δηλαδή ένα σωρό παραδείγματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Είναι δύσκολο να σπάσει κανείς τους φραγμούς αλλά εδώ και 30-40 χρόνια δεν θεώρησα ποτέ ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε και ε, δεν απογοητεύτηκα. Ε, έχουμε λοιπόν μία high level group for gender mainstreaming που καταρτίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα σωστά κριτήρια, του σωστούς δείκτες και αυτά όλα είναι θέματα στα οποία μπορεί να συμβάλλει το Ινστιτούτο και όταν έχει κανείς πίσω του ένα τόσο μακρύ αγώνα όπου έχουμε πολλές φορές κινηθεί από κοινού υπάρχει ο κίνδυνος οι γυναίκες να διαδεθούν ή να προσπαθήσει κανείς να ξεχωρίσει τις γυναίκες που εργάζονται από αυτές που όχι ή τους ακαδημαϊκούς ε, ε, τους πανεπιστημιακούς από τους, ε, τις γυναίκες που εργάζονται σε γραφείο. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ισότητα και γι' αυτό και ελπίζω και θα πρέπει με επίφαση να φροντίσουμε οι άντρες να μας ακολουθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Κυρία Μποσκουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε καλωσορίζω, Λίζη. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, παρότι παίζει ένα διαφορετικό ρόλο σήμερα στην Επιτροπή μας. Πάντως, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι υποψήφια για αυτό το φόρουμ εμπειρογνωμών. έχεις ε, μεγάλη εμπειρία, ε, δεν μπορεί κανείς να την εμφισβητήσει ε, και χαίρομαι που είσαι πρόθυμη να αναλάβεις νέες ευθύνες, νέα καθήκοντα. Έχεις μακρά πολιτική εμπειρία και θα ήθελα να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Ε, μιλάμε για ένα ρόλο συμβούλου, ρόλο εμπειρογνώμονα. Ε, αυτή είναι η θέση. Ε, μπορείς να αλλάξεις καπέλο, το πω έτσι, δηλαδή θα κληθείς να κάνεις κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτά που έκανες νωρίτερα και μπορεί να νιώσεις και απογοήτευση γιατί δεν θα είσαι πια στο φως της δημοσιότητας, στο το πω έτσι. Και η πρώτη ερώτηση προκύπτει η δεύτερη ερώτηση συγγνώμη, που θα σου θέσω προκύπτει από την πρώτη. Ε, δεδομένης της ε, οικονομικής ε, κρίση σε πολλά κράτη-μέλη διαπιστώνουμε ότι πολλοί δεν έχουν όρεξη να συζητήσουν για αυτά τα ζητήματα ισότητα των δύο φύλων. όχι, συνεπάγεται μεγάλο κόστος, κάτι τέτοιο. Ήδη δαπανώνται πολλά χρήματα για τις τράπεζες. Εμένα με ανησυχεί πάρα πολύ αυτή η τάση που σημειώνεται. Ειλικρινά πιστεύεις ότι το Ινστιτούτο με τους περιορισμένους πόρους που θα έχει θα μπορέσει να κάνει ε, κάτι σημαντικό. Και εν τη αυτή περιπτώσει ποια στρατηγική θα προτείνει στο Ινστιτούτο. Σας ευχαριστούμε. Λίζη. Μικρόφωνο παρακαλώ. ο συμβουλευτικός ρόλος ε, δίνει μεγαλύτερη ελευθερία. Δηλαδή δεν ε, ε, είμαι δεμένη με κομματικά και πολιτικά δίκτυα και πιστεύω ότι η μακροσκελή σπήρα που έχω μπορεί να έχει και αρνητικές επιπτώσεις αλλά μπορώ να αξιολογήσω πώς συνεργάζονται τα διάφορα θεσμικά όργανα. Γι' αυτό και έχω μία πείρα που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ε, έχουμε δηλαδή ε, και σε άλλα επίπεδα Ινστιτούτα τα οποία συνεργάζονται και γι' αυτό πιστεύω ότι και εδώ η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πρέπει να ακούγεται ακόμη και αν γίνει με κάποια απόσταση διότι πλέον δεν είμαι ευρωβουλευτής αλλά γνωρίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γνωρίζω και την Επιτροπή και ξέρω ότι η εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να επηρεάσει το Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και αυτό πιστεύω ότι είναι το μεγάλο προτέρημα, δηλαδή ε, να μην βρίσκεται κανείς ε, με την ευθύνη ε, μίας άμεσης εντολής αλλά να μπορέσει να συνεργαστεί χωρίς προστριβές και πιστεύω ότι έτσι θα λειτουργήσω καλύτερα και ούτως ή άλλως έχω μεγάλο στομάχι διότι διαφορετικά δεν θα είχα επιμείνει τόσα χρόνια στον τομέα της πολιτικής ισότητας των φύλων. Εάν λοιπόν κάποιος λίγο αποστασιοποιηθεί και κάνει ένα απολογισμό τι έχουμε πετύχει από όταν είμαι στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δηλαδή, ε, ε, εάν έχω δουλέψει πάνω από 20 χρόνια στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, πρέπει να πω ότι ο απολογισμός μου είναι θετικός. Έχουμε πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες πλέον ορίζουν την τύχη τους. Δεν έχουμε πετύχει τα πάντα, πολλά ακόμη πρέπει να γίνουν, αλλά οι αδερφές μας μόνο πριν από 100 χρόνια άρχισαν να ψηφίζουν. Οπότε από αυτού νομίζω ότι έχουμε κυριεύσει ε, τα κοινοβούλια πρέπει όμως τώρα να επηρεάσουμε την κοινωνία κατά τέτοιον τρόπο ώστε ε, οι άντρες και οι γυναίκες να μπορούν να αναπτύσσονται χωρίς να αποτελέσει μήλον της έριδος το φύλλο. Ε, θα ήθελα λοιπόν να συμβάλλω στις προσπάθειες αυτές και εδώ μπορώ να βοηθήσω κι εγώ διότι παρόλες τις αποτυχίες πιστεύω ότι έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο και τώρα ε, στην Ευρώπη ο ρόλος της γυναίκας είναι πολύ πιο θετικός από ό,τι σε, σε άλλα μέρη του κόσμου και ε, πιστεύω ότι γι' αυτό και ο πλούτος των εμπειριών μου μπορεί να βοηθήσει τις ε, γυναίκες με μεγαλύτερη αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε κυρία Γκρένερ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι έχεις αμύωτη δέσμευση και αφοσίωση ε, βλέπω πόσο μακρο, μακρόπνοα βλέπεις ε, το ρόλο σου. Ε, ορισμένες φορές δεχόμαστε χτυπήματα, αλλά συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας. Είχα σκεφτεί να σε ρωτήσω ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες για το Ινστιτούτο, αλλά έκανες τόσο σαφή παρουσίαση που δεν χρειάστηκε, αναφέρθηκε στις τομείς που κατά τη γνώμη σου είναι σημαντικότεροι δεδομένης και της συγκυρίας. Ε, έδωσες ε, σαφείς απαντήσεις σχετικά με τις προτεραιότητές σου. Οπότε, ε, εξ ονόματος της Επιτροπής, σε ευχαριστώ ενθέρμως για την παρουσία σου. Ε, και για, την, για τις αφέστατες ε, απαντήσεις που μας έδωσες. Καλή επιτυχία. Έλειψες σε πολλούς από μας εδώ στην Επιτροπή. Πάντως καλή επιτυχία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα εδώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Μανταριάγκα Αμπεραστούρη ε, που έχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Βασκικού Ινστιτούτου για τις Γυναίκες ε, στην Ισπανία. Καλωσορίσατε. Ε, παρακαλείστε θα μας κάνετε μια δεκάλεπτη περίπου παρουσίαση ε, για να μας μιλήσετε για την εμπειρία που έχετε στον τομέα και να μας ε, πείτε ακριβώς σε τι θα μπορούσατε να βοηθήσετε, τι θα μπορούσατε να συνεισφέρετε στο φόρουμ των εμπειρογνωμόνων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής, κυρίως για αυτή την πρόσκληση. Ο καλύτερος τρόπος ε, να προσπίσω την υποψηφιότητά μου ως ε, υποψήφια είναι να σας παρουσιάσω τις δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην ε, επίτευξη των στόχων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Υπήρξα Γενικός Γραμματέας του Βασκικού Ινστιτούτου τα τελευταία τέσσερα χρόνια και ενδιαφέρομαι να μάθω και να αναπτύξω καινούριου τομεί. Έχετε το βιογραφικό μου σημείωμα με ενδελεχεί πληροφορίε για την πείρα μου και θα ήθελα απλώ να επισημάνω κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. As executive director... Ως ε, Γενική Διευθύντρια ήμουν υπεύθυνη για την ε, διοίκηση του Ινστιτούτου, κυρίως ε, την διοίκηση του προσωπικού και τη διοίκηση του προπολογισμού συντόνισα τις εργασίες μεταξύ των διαφόρων ομάδων. Ε, πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκα με πολιτικά, τεχνικά και κοινωνικά θέματα και είμαι επίσης ε, δικηγόρος ειδική σε θέματα βίας κατά των γυναικών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχω πείρα ως ε, εκλεγμένο μέλος της ε, οργάνωσης δήμων και κοινοτήτων και περιφερειών της Ευρώπης. Θα ήθελα να επισημάνω επτά προτεραιότητες, τις οποίες έχω προασπίσει στο ε, Βασικό Ινστιτούτο και σκοπεύω να ε, προωθήσω και στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Πρώτον, gender mainstreaming και η ένταξη της πτυχής του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικής. Ε, ισότητα για τους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα. Διαθεσμικό συντονισμός, συντονισμός μεταξύ των διαφόρων φορέων σε θέματα βίας κατά των γυναικών, δημιουργία ενός ε, γραφείου ισότητας, έκτον, δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γυναικών και έβδομον, προώθηση πολιτικών ισότητας που απευθύνονται σε άνδρες. Να τα αναπτύξω πιο αναλυτικά. Η ένταξη της διάταξης του φίλου. Χρειαζόμαστε πολιτικές για να διαπιστώσουμε κατά πόσον ε, οι πολιτικές ισότητας εφαρμόζονται και αν έχει θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία. Αν όχι, θα πρέπει να έχουμε τα σωστά διορθωτικά μέτρα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μέσα για τα ε, για τους δημόσιους θεσμούς και αυτό θα πρέπει να αποτελέσει ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα του Φύλου διότι θα είναι αυτό το οποίο θα ασχοληθεί με την ισότητα των φύλων. Θα μπορέσει επίσης να ομογενοποιήσει τη συλλογή δεδομένων και τα στατιστικά στοιχεία της κάθε χώρας. Δεύτερον, κατάρτιση. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο θα πρέπει να δίνει συμβουλές και να προάγει τις ε, ισότητα για τους ε, δημοσίους υπαλλήλους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως απαραίτητο μέτρο για την ε, ενσωμάτωση της πτυχής του φύλου στις δημόσιες πολιτικές. Τρίτον, διαθεσμικός συντονισμός σε θέματα συντονισμού μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα μόνο αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων ακολουθώντας τους ίδιους κανόνες. Και αυτό αποτελεί ευθύνη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές πραγματικότητες που ισχύουν στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτήν την έννοια θα ήταν πολύ χρήσιμο να μπορέσουμε να συνεργαστούμε με την ε, Επιτροπή των Εκλεγμένων Γυναικών στους Δήμους και Περιφέρειες της Ευρώπης, η οποία ασχολείται τα τελευταία 25 χρόνια με τον τομέα αυτό. Το τελευταίο της επίτευγμα είναι η Ευρωπαϊκή Επιστολή για την Ισότητα. Τέταρτον, ο διαθεσμικός συντονισμός ε, για τη βία αφορά τόσο την ε, ε, πάταξη της βίας αλλά και την ε, φροντίδα των θυμάτων βίας. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιτείνονται από τη βία και θα πρέπει να μπορέσουμε να συνεργαστούμε για να σταματήσει η βία. Επίσης, θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκτυα, δίκτυα τα οποία θα περιλαμβάνουν μικτά τα Ινστιτούτα, ε, ενώσεις γυναικών και ούτε καθεξής. Αυτό θα μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε τη βία κατά των γυναικών και να βελτιώσουμε την φροντίδα που προσφέρεται σε όλα τα θύματα ε, βία στο σπίτι ανά την Ευρώπη. Πέμπτον, το Βασικό Γραφείο άμυνας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος δημιουργήθηκε το 2006 is the defense of Στόχος είναι η προάσπιση ανδρών και γυναικών ε, όταν είναι θύματα διάκρισης ε, σε θέματα φύλου. Είχαμε μέχρι τώρα τα θέματα διακρίσεων ε, κατά των γυναικών στον ιδιωτικό τομέα. Ε, θα πρέπει να συντονιστούν οι διάφοροι φορείς που υπάρχουν στα κράτη-μέλη και θα μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί το Ινστιτούτο ως παρατηρητήριο για τις διαφορετικές περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε στις ευρωπαϊκές χώρες. Έκτον, έναν Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γυναικών, ένα ε, φορέα συμμετοχής των γυναικών. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο θα πρέπει να προάγει και να προτείνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Γυναικών, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ε, γνωρίζουμε πώς προχωρεί το κίνημα των γυναικών και να έχουμε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το οποίο θα μπορέσει να βοηθήσει και τη συμμετοχή των γυναικών στον ευρωπαϊκό τομέα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να ε, απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλο, θα ήθελα να σα πω ότι αναγνωρίζω ότι το γεγονό ότι η αποτελεσματική ισότητα δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν προχωρήσουν και οι άνδρες από κοινού με τι γυναίκες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το 50% τη κοινωνία μα να μείνει πίσω. Θα πρέπει λοιπόν να πράγουμε και πολιτικέ για του άνδρες, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ενθαρρύνουμε και του άνδρες και τι γυναίκε, να συνεργαστούν και να ακολουθήσουν τις ίδιες ε, άγουσες στην αναζήτηση της ισότητας. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ινστιτούτο θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της συνεργασίας με τους άνδρες και να τους ενσωματώσει στις δημόσιες πολιτικές για την ισότητα που αναπτύσσονται στην Ευρώπη. Εν κατακλείδη, κανένα από αυτά δεν μπορούμε να τα επιτύχουμε χωρίς την πολιτική υποστήριξη και τη δέσμευση των μελών αυτής της Επιτροπής. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σε 10 λεπτά. Αν όμω κάποιο από εσά ε, θέλει να μου θέσει κάποια ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις ε, των μελών της Επιτροπής μας. Παρακαλώ, η κυρία Κορνέλη. Ναι, σας ευχαριστώ για την ε, παρουσίασή σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η απαρίθμηση των στοιχείων που θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Συμφωνώ. Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για την οργάνωση της οποίας είστε Γενική Γραμματέας. Γιατί λέει ότι ε, απευθύνεται στους ε, δήμους της χώρας των Βάσκων. Ασχολείστε λοιπόν με θέματα ισότητας των φύλων ε, σε τοπικό επίπεδο ή ε, εξετάζετε και τις ευρωπαϊκές πτυχές. Τι εμπειρογνωμοσύνη λοιπόν έχετε σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή έρευνα σε θέματα ισότητας των φύλων. Ευχαριστώ κύριε Κορνελίσεν. Παρακαλώ. Η δουλειά μου στο Βασκικό Ινστιτούτο για τις Γυναίκες Το Βασκικό Ινστιτούτο πρέπει να σας πω ότι ήταν πάντα πρωτοπόρο σε πολιτικές ισότητες και κατά κάποιο τρόπο αναγνωρίστηκε πάντα το έργο του και εντός της Ισπανίας αλλά και στην Ευρώπη σε άλλα Ινστιτούτα, σε άλλους οργανισμούς ε, και σε άλλες οργανώσεις γυναικών ε, στην Ευρώπη. Ε, η συνεργασία τώρα με τους Δήμους. Εγώ θα πρέπει να κάνω ένα διαχωρισμό εδώ. Αφενός εργάστηκα στην Επιτροπή Γυναικών του Συμβουλίου Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης ως ε, δήμαρχος μιας περιοχής της οποίας ήμουν όταν πριν έργα στο Βασικό Ινστιτούτο. Επειδή όμως γνωρίζω και τι δύο περιπτώσεις, δηλαδή και πώ λειτουργούν τα κυβερνητικά θέματα, όπως λειτουργούν και οι Δήμοι, ε, Πρέπει να σας πω ότι έχω και την πείρα στο βασικό Ινστιτούτο και η συνεργασία με τους Δήμους είναι πολύ σημαντική σε αυτή την περίπτωση. Διότι οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι πιο κοντά στον λαό, αυτοί που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά σε ποιον πληθυσμό απευθύνουν τις πολιτικές τους, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά αν υπάρχουν αποτελέσματα στις πολιτικές ή στις δράσεις ε, που εφαρμόζουν οι Δήμοι και αυτό που πάντα θεωρούσαμε δεδομένο είναι ότι οι οργανισμοί ισότητα σε αυτή την περίπτωση ε, τουλάχιστον στη χώρα των Βάσκων έπρεπε να είναι σε πλήρη συνεργασία με τους Δήμους. Γι' αυτό ακριβώς και το 2004 δημιουργήθηκε ένα δίκτυο βασικών ε, δήμων ε, για την καταπολέμηση της βίας και την ισότητα των φύλων, στην οποία συνεργαζόταν και το Βασικό Ινστιτούτο για τη Γυναίκα και ε, ο οργανισμός ΕΟΥΜΠΕΛ που συμμετέχει και στην Επιτροπή Περιφερειών και Δήμων της Ευρώπης. Η συνεργασία αυτή ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Καταφέραμε λίγο πολύ το 80% του πληθυσμού της χώρας των Βάσκων να ζει σε ένα δήμο όπου υπάρχει ένα πρόγραμμα ισότητας ε, σε πρακτική εφαρμογή, δεν είναι κάτι το οποίο απλά έχει εκπονηθεί, αλλά έχουν ε, δαπανηθεί και τα κονδύλια και το προσωπικό προκειμένου να προχωρήσουν αυτά τα προγράμματα. Υπάρχουν πρωτόκολλα ε, υλοποίησης μέσω αυτού του δικτύου προκειμένου όλοι οι δήμοι, σε αυτή την περίπτωση της χώρας των Βάσκων, να διαθέτουν τα ίδια μέσα αλλά και τους ίδιους στόχους όπως και τα σχέδια, διότι τα σχέδια για την ισότητα των Δήμων σε κάποιο βαθμό υπόκεινται και σε ένα ε, σχέδιο πλαίσιο το οποίο εκπονεί το Βασκικό Ινστιτούτο για τη Γυναίκα και ο τελικός μας στόχος είναι όλοι οι Δήμοι και όλες οι γυναίκες των Δήμων της χώρας των Βάσκων να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις τις οποίες θα μπορούν να ασκήσουν και το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και τους άνδρες τώρα. Γι' αυτό ακριβώς πρότεινα να υπάρχει μια άμεση συνεργασία μεταξύ του Ινστιτούτου ε, για την ισότητα των φύλων και τους Δήμους και τις περιφέρειες, διότι εγώ εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια στον τομέα αυτό και πραγματικά οι Δήμοι πρέπει να σας πω ότι είναι αυτοί που γνωρίζουν την πραγματικότητα και την κατάσταση ε, των γυναικών της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πάνοβα. Thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. με εντυπωσιάζει όχι μόνο η δουλειά σας αλλά και η προσέγγισή σας διότι αυτό που μας παρουσιάσατε μοιάζει με σχέδιο εργασίας και αυτό είναι αυτό το οποίο αναζητούμε. Γι' αυτό άλλωστε και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι έχετε μια εκτελεστική προσέγγιση των πραγμάτων. Αυτό που με εντυπωσίασε επίσης είναι τα σημεία 2, 4 και 7. Το 7 αφορούσε στους άνδρες και Ο συνάδελφος από την Ελλάδα εδώ έθεσε ένα θέμα και λέει ότι όχι μόνο δεν είναι, είναι ο μόνος άνδρας, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που προτείνεται. Θα ήθελα να σας θέσω δύο ερωτήσεις. Για τα σημεία 2 και 4 νομίζω στα οποία αναφερθήκατε. από τι θα αποτελείται αυτή η κατάρτιση για την ισότητα στο δημόσιο τομέα, γιατί αυτό είναι κάτι πολύ καινοτόμο που μας προτείνεται και επίσης η τέταρτη παρατήρησή σας, τι προτάσεις έχετε για την φροντίδα των θυμάτων βίας και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου, διότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ε, θα συζητήσει η Επιτροπή μας, θα παρουσιάσουμε και σχετική προφορική ερώτηση συζητάμε πάρα πολύ για τη βία, αλλά δεν συζητάμε ποτέ τη φροντίδα των θυμάτων ε, βίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Επειδή εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια σε έναν ε, οργανισμό ισότητας, και προσπάθειά μας είναι οι δημόσιες πολιτικές να περιλαμβάνουν και τη διάσταση του φύλου, ε, αντιληφθήκαμε και όχι μόνο το αντιληφθήκαμε αλλά και οι ίδιοι υπάλληλοι των ε, διοικήσεων ήθελαν να υπάρχει και σχετική κατάρτιση σε θέματα φύλου για να μπορέσουν να κάνουν και τη δουλειά τους. Βέβαια δεν κάνουν όλοι οι υπάλληλοι της διοίκησης την ίδια δουλειά, αλλά εγώ προτείνω, γιατί αυτή είναι και η πείρα που έχω από τη χώρα των Βάσκων και λειτουργεί πάρα πολύ καλά το σύστημα, η κατάρτιση σε θέματα ισότητας να είναι για όλη τη διοίκηση. Ε, βέβαια, ο καθένας και η κάθε μία ανάλογα με αυτό που πρέπει να κάνει. Μπορεί κάποιος ε, να πρέπει να ε, εκπονήσει κανόνες και θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει πολύ καλά πώς ε, εντάσσεται η διάσταση του φίλου στις τομεακές πολιτικές. Θα πρέπει να γνωρίζει δεδομένα, να έχει στατιστικά στοιχεία, να ξέρει ε, σε ποιες περιπτώσεις συμβαίνει τι, τι επιπτώσεις έχουν όλες αυτές οι δράσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες. Θα πρέπει να μπορεί να αναλύσει αυτά τα δεδομένα και αυτά απαιτούν μία κατάρτιση. Κανένας δεν μαθαίνει για την ισότητα εάν δεν του τη διδάξουν και αν δεν βρεθεί ενώπιον πολύ συγκεκριμένων δεδομένων το οποίο το επιτρέπουν να διαπιστώσει γιατί ακριβώς μιλάμε όταν μιλάμε για ενσωμάτωση τη διάστασης του φύλου. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι, άνδρες και γυναίκες που θεωρούν ότι οι κανόνες που εκπονούν είναι ουδέτεροι. Αν λοιπόν κάποιος δεν τους διευκρινίσει ε, πού υπάρχουν οι διαφορές στους κανόνες δεν το διαπιστώνουν και δεν το διαπιστώνουν διότι δεν υπάρχει η κατάλληλη εκπαίδευση για να γνωρίζουν ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες ε, που μπορεί να έχουν οι πολιτικές σε άνδρες και γυναίκες. Γι' αυτό ακριβώς Είπαμε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά πώς ενσηματώνεται η διάσταση του φύλου στους κανόνες. Επίσης υπάρχουν υπάλληλοι σε διοικήσεις που θα πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή προγράμματα δράσης και μάλιστα σε πολύ διαφορετικούς τομείς. Μπορεί να γνωρίζουν πολύ καλά τον τομέα, για παράδειγμα τον τομέα της βιομηχανίας, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να μην γνωρίζουν πώς μπορεί να υπάρχει ένα ε, θετικό πρόγραμμα δράσης, πώς μπορούν να ενσωματίσουν τη διάσταση του φύλου στα όσα ετοιμάζουν για την τομεακή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουν και την ανάλογη εκπαίδευση ε, για το θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να καταρτίζεται το προσωπικό προκειμένου να ε, χρησιμοποιούν ορολογία ε, όπου δεν θα υπάρχουν διάκριση. Πολλές φορές ε, τα διοικητικά έγγραφα δεν ε, είναι ανάλογα ευαισθητοποιημένα. Είναι πάντα σε γένος αρσενικό, διότι θεωρούν ότι το αρσενικό γένος ε, αφορά και άνδρες και γυναίκες. Ιστορικώς έτσι γινόταν. Αλλά κατά κάποιο τρόπο θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε είτε όρους οι οποίοι θα είναι ουδέτεροι και δεν θα απευθύνονται μόνο σε άνδρες και γυναίκες, αλλά θα απευθύνονται γενικότερα στους πολίτες, ή να χρησιμοποιείται ξεχωριστά το αρσενικό και το θηλυκό γένος, μπορεί βέβαια τα κείμενα έτσι να γίνονται μεγαλύτερα και να περιλαμβάνουν ίσως και ε, στοιχεία που μπορεί να αποτελούν πρόβλημα. Θα πρέπει όμως να γίνεται πράγματα στους τομείς αυτές και θα πρέπει να υπάρχει και μια γενική κατάρτιση ως προς την ορολογία, τι είναι ο φεμινισμός, την ισότητα, πράγματα τα οποία είναι βασικά, αλλά καλό θα ήταν να τα γνωρίζουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι σε επίπεδο διοικητικό, τεχνικό αλλά και πολιτική και ε, πολιτική που ε, είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή αυτών των ε, ε διοικήσεων διότι πολλές φορές πρέπει να κάνουν πολιτική, να παράξουν πολιτική και δεν ξέρουν τα θέματα της ισότητας των φίλων. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα για τη δεύτερη ερώτηση που μου θέσατε. για τον ε, συντονισμό σε θέματα ε, φροντίδας ε, θυμάτων ε, βία στο σπίτι, ο συντονισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλα τα θεσμικά όργανα τα οποία συνεργάζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα με ε, γυναίκες οι οποίοι είναι θύματα βίας από άνδρες θα πρέπει να συνεργάζονται και να έχουμε την ίδια γραμμή πλεύσης. Τι προτείνω. Προτείνω να συνεργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να υπάρχει ένα όργανο συντονισμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου και των άλλων Ινστιτούτων γυναικών που υπάρχουν στις υπόλοιπε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να γνωρίζουμε τι μέτρα και τι ε, φροντίδα λαμβάνουν σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης οι γυναίκες οι οποίες είναι θύματα βίας. Να καθορίσουμε πρωτόκολλα δράσης προκειμένου να εφαρμόζονται για γυναίκες που είναι θύματα βίας, να γνωρίζουμε τι ε, υπηρεσίες υγείας υπάρχουν, τι δικαστικά βήματα πρέπει να λάβουν, τι πρέπει να κάνει η αστυνομία για μια γυναίκα η οποία υπήρξε θύμα βία στο σπίτι. Εμείς στη χώρα των Βάσκων από το 2001 έχουμε μια διαθεσμική συνεργασία ε, συμφωνία συγγνώμη, για τη συνεργασία για όλες αυτές τις πολιτικές και υπάρχει ένα πρωτόκολλο δράσης το οποίο τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μόλις υπάρξει επίθεση σε μια γυναίκα στη χώρα των Βάσκων. Ε, λειτουργεί 8 χρόνια. Ε, όλοι όσοι συμμετέχουν το αξιολογούν θετικά ε, και είναι αλήθεια ότι ακόμα και οι ίδιες οι γυναίκες οι οποίες υπήρξαν θύματα αξιολογούν θετικά τα όσα έχουν γίνει για αυτές. Όλα λοιπόν όσα αφορούν ε, θέματα συνεργασία μεταξύ Ινστιτούτων, κυρίω συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι είναι πολύ πιο δύσκολο για ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο να έχει άμεση επαφή με γυναίκα στήματα. Η άμεση συνεργασία λοιπόν με μη κυβερνητικού οργανισμού που τόσα χρόνια ε, ήταν ουσιαστικά η φωνή και αυτοί οι, οποίες, ε, οι οποίοι φρόντισαν γυναίκε στήματα. Είναι αυτοί που γνωρίζουν την κατάστασή του και γνωρίζουν και τι πρέπει να κάνουν τα διάφορα Ινστιτούτα. Θεωρώ ότι αυτά είναι από τα βασικά σημεία τα οποία θα πρέπει ε, να φροντίσει το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε η κυρία Μποσκότ και η κυρία Μπιλμπάου μετά. Ε, καλωσορίσατε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. απαριθμίσατε τους στόχους σας, πράγματα που θέλετε να υλοποιήσετε. Δυστυχώς ε, το Ινστιτούτο αυτό δεν θα έχει επαρκείς πόρους ε, στη διάθεσή του, άρα πρέπει να περιοριστείτε κάποιους Ποιες είναι οι ύψιστες προτεραιότητες του προγραμματός σας. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, χωρίς να σας μιλήσω για τις δικές μου προτεραιότητες. Ε, ξέρετε, λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε δώσει εκατομμύρια στις τράπεζες, αλλά για την άδεια μητρότητες ε, ή για άλλα ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα των δύο φύλων, όλα κρίνονται υπερβολικά ακριβά και δεν χρηματοδοτούνται. Ε, είναι δυσχερής η περίοδος λοιπόν για τον τομέα που μας απασχολεί. Εάν ε, επιλεχθείτε, ε, για, αν διοριστείτε στο Ινστιτούτο, λοιπόν, ποια είναι η στρατηγική που θα προωθήσετε, ούτως ώστε να γίνει πιο επίκαιρο το θέμα της ισότητας ε, των δύο φύλων. Παρακαλώ. Αν έπρεπε να διαλέξω μία προτεραιότητα, κάτι το οποίο είναι δύσκολο, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η διαθεσμική συνεργασία στο κάτω-κάτω της γραφής υπάρχουν και άλλα Ινστιτούτα που εργάζονται για θέματα ισότητας των φύλων σε, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Επομένως, ένα Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο αυτό που θα πρέπει να κάνει πρωτίστως είναι να συντονίσει όλο το έργο των Ινστιτούτων ε, της γυναίκας για να γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Αν πρέπει να επιλέξω μόνο ένα. Εγώ βέβαια προφανώς θεωρώ ότι όσο μικρό και αν είναι αυτό το Ινστιτούτο θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ φιλόδοξοι και οι στόχοι θα πρέπει να είναι σημαντικοί. Και εγώ εργάστηκα σε ένα πάρα πολύ μικρό Ινστιτούτο, αλλά πάρα πολλές φορές η διάθεση να κάνουμε πράγματα και ε, η αγάπη για τη δουλειά ε, μπορεί να μας ε, βοηθήσει πολύ περισσότερο από τα μέσα. Ξέρουμε ότι η Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπάρχουν πάρα πολλές χώρες που διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ των, αλλά αν πρέπει να διαλέξω ένα καθήκον, αυτό θα ήταν η διαθεσμική συνεργασία μεταξύ των Ινστιτούτων. Ε, και το δεύτερο, για να μην μακρηγορήσω, το θέμα της οικονομικής κρίσης. Δυστυχώς, όταν δεν υπήρχε οικονομική κρίση, πάλι δεν είχαμε και πάρα πολλά χρήματα για την ισότητα. Η ισότητα πάντα ήταν η πολιτική ε, των φτωχών. Υπάρχουν πάντα πολιτικές πολύ πιο σημαντικές Εάν λοιπόν πριν ε, που ήταν πολύ καλή οικονομική κατάσταση δεν ήταν σημαντικό ο προπολογισμό που διατίθεταν για την ε, ε, ισότητα, φαντάζομαι ότι τώρα θα είναι πολύ λιγότερο. Αλλά εγώ αυτό δεν θα το ρίξω στην οικονομική κρίση. Ε, πρέπει να γίνει πολύ σημαντική δουλειά από πλευρά Ινστιτούτο, πρέπει να κάνει πολύ σημαντική δουλειά και η Επιτροπή σα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Θα πρέπει στην ατζέντα των πολιτικών τη Ευρώπη να υπάρχει το γεγονός ότι η ισότητα είναι πολύ σημαντική. Το ξέρω ότι υπάρχουν πολύ πιεστικά θέματα, πολύ πιο πιεστικά, αλλά το θέμα της ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα θέμα το οποίο ε, αν δεν πρέπει να βρίσκεται στην πρώτη θέση θα πρέπει τουλάχιστον να βρίσκεται στη δεύτερη θέση των προγραμμάτων ε, των ευρωπαϊκών χωρών. Λοιπόν, πάει λίγο πιο πάνω στην ατζέντα θα είχε πολύ περισσότερα χρήματα. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα, με ή χωρίς κρίση. Εγώ λοιπόν δεν θα ε, ρίξω το φταίξιμο στην κρίση, διότι δυστυχώς ήταν πάντα μία από τις φτωχές πολιτικές. Να δούμε αν θα αλλάξουν τα πράγματα. Ως προς τις στρατηγικές, δεν θυμάμαι πώς τέθηκε η ερώτηση. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε wat voor strategie zou u adviseren? Ναι, η στρατηγική σας σας ρώτησα. Ποια στρατηγική μπορείτε να εισηγηθείτε στο Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων, ούτω ώστε να γίνει επίκαιρο το θέμα, να έχει μεγαλύτερη διασημότητα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική ευαισθητοποίηση. Η κοινωνία πολλές φορές ε, ζητά συγκεκριμένη δουλειά. Όταν η κοινωνία ζητά ε, ισότητα, οι πολιτικοί δεν έχουν άλλη λύση από το να ε, βρουν μία λύση για αυτό που τους ζητάνε. Εάν λοιπόν η κοινωνία είναι ευαισθητοποιημένη και πρέπει εδώ να γίνει και μία δουλειά ευαισθητική, ίσως πολύ σημαντική σε θέματα ισότητας της κοινωνίας μας, ε, και τότε μόνο θα ζητήσουν από τους πολιτικούς τους, άνδρες και γυναίκες, να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να αλλάξει καταρχάς η νοοτροπία και κατόπιν οι πολιτικές ε, σε θέματα ισότητας των φύλων και να ενσωματωθεί η ισότητα των φύλων όπως κάθε εγκάρσιο θέμα στις θεμαϊκές πολιτικές όπως έγινε με το περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλο θέμα. Το πρώτο όμως είναι ότι η κοινωνία θα πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ισότητα και πόσο σημαντική είναι η δουλειά για την ισότητα και να απαιτήσει από τους πολιτικούς τις άνδρες και γυναίκες να εργαστούν από αυτού. Ωραία, τώρα ας ακούσουμε την κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και την κυρία Μανταριάγκα. Καταρχάς γιατί είσαστε πολύ συγκεκριμένοι και γιατί μας δώσετε μια πολύ σαφή ιδέα για το τι σημαίνει για σας ένα Ινστιτούτο, ένα πρακτικό Ινστιτούτο με συγκεκριμένα μέσα και με άμεσες δράσεις. Σα έθεσαν αρκετέ ερωτήσει και μου απαντήσατε κάποια ερωτηματικά. Μιλήσατε για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα στο οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι άνδρε. Η ερώτησή μου το Βασικό Ινστιτούτο για τη Γυναίκα, το Εμμακούντε, πότε θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντική η ενσωμάτωση των ανδρών. Τι συνέβη, έχετε συγκεκριμένη εμπειρία από αυτού και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Και δεύτερον, όσον αφορά στη συμμετοχή των γυναικών, στα βασικά Ινστιτούτα υπάρχει σημαντική παρουσία γυναικών, κυρίω τα τελευταία δύο χρόνια. Θα ήθελα να γνωρίζω λοιπόν ε, σε τι οφείλεται, τι μέτρα ε, προώθηση του Ινστιτούτου και πώς το αντιλήφθηκαν αυτό και όσο ο πολιτικός αλλά όσο και ο κοινωνικός ε, χώρος, η πραγματικότητα. Έχετε συνεργαστεί με μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι αποτέλεσμα υπήρχε εκεί. Υπάρχουν ε, κυρώσεις, μέτρα που αφορούν σε κυρώσεις ως προς τις εικόνες και την ορολογία, το λεξιλόγιο που διαβιβάζεται. Έχετε συνεργαστεί με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου εκεί υπάρχει πολύ μεγαλύτερη έλλειψη από ό,τι στο δημόσιο τομέα όσον αφορά σε θέματα ισότητας. Και τέλος αναφερθήκατε σε ένα καινοτόμο Ινστιτούτο, το, αυτό το Ινστιτούτο Άμυνας ε, το οποίο αναφέρεται. Τι ακριβώς κάνει αυτό το Ινστιτούτο Άμυνας και πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτό το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Να τα δούμε τμήματικά. Ως προς τη συμμετοχή των ανδρών. Μετά από πολλά χρόνια δημιουργίας πολιτικών ισότητας, αντιληφθήκαμε ότι οι πολιτικές ισότητας ε, που γίνονται από τα Ινστιτούτα και από τα θεσμικά όργανα δεν φτάνουν στους άνδρες. Δεν συμμετείχαν στις δραστηριότητες, όσο ενδιαφέρον και αν ήταν, όσο τομεακές και αν ήταν, η συμμετοχή των ανδρών λοιπόν σε όλα όσα είχαν σχέση με ισότητα των φύλων ήταν ελάχιστη και διαπιστώναμε ότι οι γυναίκες προχωρούσαν σε πάρα πολλά θέματα και οι άνδρες δεν είχαν εξελιχθεί αναλόγως ώστε να βρίσκονται επίσης όρις με τις γυναίκες. Γι' αυτό λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε ένα βήμα με κάποιο τρόπο. Το 2001 από το Ινστιτούτο έγινε το πρώτο συνέδριο για τη συμμετοχή των ανδρών και το 2007 επανήλθε το θέμα της συμμετοχής των ανδρών και επανήλθε από πλευράς Ινστιτούτου κυρίως, διότι τότε ο πρόεδρος ε, της κυβέρνησης, ο λέντακαρι ο Ιμπαρέτσε, ενδιαφερόταν ιδιαίτερα ως άνδρας να υπάρχει κάποια ε, πρωτοβουλία της κυβέρνησης που θα απευθύνεται στους Βάσκους άνδρες. Γι' αυτό ακριβώ και σχεδιάστηκε αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ονομάστηκε Βυσόντους και θέμα ε, είχε την ισότητα ως προς τον άνδρα. Και ποιος ήταν ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας. Ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή των ανδρών σε θέματα ισότητας και να υπάρχει και μια αλλαγή από πλευράς ε, κοινωνίας ε, ως προς την οτροπία της. Τι κάναμε. Κάναμε μια σειρά από μέτρα τα οποία βασίζονταν σε τρεις πυλώνες, την ευαισθητοποίηση, την κατάρτιση και τη συμφιλίωση και συνυπευθυνότητα. Σε θέματα ευαισθητοποίησης ε, ξεκίνησαν κάποιες συγκεκριμένες διαφημιστικές εκστρατείες ε, οι οποίες σε κάποιο βαθμό προσπαθούσαν να δούμε και τι άνδρες αρέσουν στις γυναίκες, τι ζητάμε από τους άνδρε, από του νέου αυτού άνδρες που θέλουμε να είναι συντροφοί μα σε αυτό το καθήκον ε, κάναμε διαφημιστικές εκστρατείες, έγιναν και κάποια ε, άλλα θέματα κατάρτισης. Υπήρξε και κατάρτιση διότι σε κάποιο βαθμό διαπιστώσαμε ότι πολλές φορές οι άνδρες δεν ξέρουν τι είναι αυτό που τους ζητάμε να αλλάξουν. Ε, ήθελα να ξέρουν ποιο είναι το νέο μοντέλο του αρενοπού άντρα, πώς μπορούμε να σπάσουμε τα ιστορικά στερεότυπα και να τους δώσουμε και κάποιους τρόπους για να το κάνουν αυτό. Και φυσικά το να προσέχουν, ε, να βοηθούν στο σπίτι, να γνωρίζουν λίγο τι ακριβώς χάνουν, επειδή ακριβώς δεν ε, συμμετέχουν σε αυτό το τομέα. Υπήρχε πολύ μεγάλη επιτυχία ε, και είμαστε στο 2009, βλέπουμε τι επιτυχία ε, υπάρχει και νομίζω ότι αυτό μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε χώρο της Ευρώπης και θα μπορούσε να το προωθήσει και το Ινστιτούτο. Πρέπει να ολοκληρώσω το ξέρω. προ τη συμμετοχή των γυναικών, να σα πω ότι η δική μα. ε, πρωτοβουλία ήταν το σχέδιο νόμου για τη συμμετοχή των γυναικών που είχε την, ως αποτέλεσμα την, την ε, συμμετοχή των γυναικών που θα μπορούσαν να έχουν άμεσες επιπτώσεις σε συζήτηση με τις κυβερνήσεις και τις διοικήσεις για τις πολιτικές για τις γυναίκες και να μην γίνεται πολιτική στο περιθώριο των γυναικών. Πρέπει να σταματήσω, ε. Με συγχωρείτε. Εξ ονόματος ε, της Επιτροπής σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσίασή σας. Ε, έχετε σαφείς προτεραιότητες και δώσατε και σαφείς απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Καλωσορίζουμε την κυρία Βίλεμ Ρούιγκροκ από την Ολλανδία. Είναι ε, σύμβουλος πολιτικής για την ε, ηλεκτρονική ποιότητα ε, και συνεργάζεται με το Κέντρο Γνώσεων για τα θέματα φύλου και διαφορετικότητας. Ε, καλωσορίσατε. Ε, έχετε 10 λεπτά για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις που θα θέλουμε να σας κάνουμε στη συνέχεια. Σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι η τελευταία και ελπίζω ότι έχετε ακόμη τη δυνατότητα και το σθένος να με ακούτε. Ευχαριστώ που με περιμένατε. Τώρα είμαι εδώ, δυναμικότατη και θα κάνω την παρουσίασή μου Ολλανδικά. Κυρία Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη τιμή για μένα να είμαι εδώ σήμερα και πρέπει να σας πω ότι ήταν μεγάλη έκπληξη το ότι με καλέσατε. προχθές ε, πρόκειτο να πάω στη Ζάμπια για ένα σημαντικό πρόγραμμα και ε, μου ζήτησαν να στείλω το βιογραφικό μου ε, γιατί μπορεί να θεωρόμουν σαν υποψήφιος εμπειρογνώμων για το Ινστιτούτο Ισότητος ε, δεν, σας, ε, δεν ήταν πολύ πλήρες το βιογραφικό αυτό. Δεν σας είπα το 80 είχα ε, συνεργαστεί με ευρωβουλευτές σαν τη Σιμών Βέιλ ότι η δεκαετία του 90 κατήρτιζα μία έκθεση για το τι γινόταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάθε τρίμηνο. Επίσης ότι έχω απαντήσει σε ερωτήσεις του Κογκρέσου όσον αφορά τις οδηγίες για την ισότητα των φύλων. Πολλά στοιχεία δεν έχουν περιληφθεί λοιπόν στο βιογραφικό μου, αλλά ίσως με ζητήσατε, μου ζήσατε να έρθω διότι θεωρήσατε ότι ήταν ενδιαφέρον το βιογραφικό μου. Ορισμένοι ίσως με γνωρίζετε γιατί έχω έρθει σαν εμπειρογνώμων πολλές φορές στην Επιτροπή σας. Ευχαρίστως θα θα αναλάβω τη θέση αυτή παρόλο που υπάρχει περιορισμένος προϋπολογισμός και μόνο τρία άτομα προσωπικό αλλά ε, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες είναι λοιπόν βασικό οι προσδοκίες αυτές να μπορέσουν να γίνουν ε, επιτεύγματα και να προωθηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο υπό τη μορφή ενός εφικτού προγράμματος. Επίσης είναι βασικό να είναι κανείς ε, εμπειρογνώμονας που να έχει καλές σχέσεις με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εστιαστούμε και να αποφύγουμε να αποτύχουμε. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε ε, καλοί εκπρόσωποι για τα δικαιώματα των γυναικών. Πρέπει λοιπόν να σας πω γιατί εγώ μπορώ να ε, έχω καλή απόδοση σε τρία θέματα. Καταρχήν, επί πολλά χρόνια έχω εμπειρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική ισότητα των φύλων εδώ και 30 χρόνια από το 79. Ήταν ε, η πρώτη χρονιά που είχαμε άμεσες ε, ε, εκλογές των Ευρωβουλευτών και τότε είχε καταρτιστεί ο προπομπός της τωρινής επιτροπής και παρακολουθούσε και τότε τα θέματα ισότητας των φύλων. Ήμουν λοιπόν παρούσα έκτοτε και ε, παρακολουθούσα τις διεθνείς εξελίξεις ε, εκ του σύνεγγης. Η Επιτροπή αυτή κατάφερε να αναπτυχθεί πολύ καλά και να περάσει διάφορες οδηγίες που υιοθετήθηκαν διαμέσου της πολιτικής διαδικασίας. Νομίζω λοιπόν ότι πετύχαμε αρκετά. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων ή τον προϋπολογισμό των φύλων, gender budgeting, πριν από 30 χρόνια ούτε είχαμε ακούσει τον όρο, ενώ τώρα είναι κάτι που είναι καθημερινό και ε, το ίδιο ισχύει και με το φόρουμ. Δεν γνωρίζω ενδεχομένως πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, αλλά ξέρω τι γίνεται στην Ευρώπη, στην Ολλανδία και όταν πρόκειται για πολιτική ε, μπόρεσα να συμμετάσχω σε διάφορα διάφορα συνέδρια, έχω πολλές επαφές, ιδίως στα νέα κράτη-μέλη, γιατί συμμετείχα σε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουμε την ευαισθητοποίηση για τις ε, νέες οργανώσεις, ε, ιδίως όσον αφορά θέματα της ισότητας των φύλων. Και έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και στην Τουρκία είναι λοιπόν πολλές οι πληροφορίες τις οποίες ε, έχω συγκεντρώσει σχετικά με την ε, καθημερινή ε, δουλειά των γυναικών. Επίσης έχω γνώσεις σε άλλα θέματα ε, κατάργησης των διακρίσεων διότι από το, τη συνθήκη του Άμστερνταμ στην Ολλανδία έχουμε το άρθρο 13 ε, είναι ε, μία πλατφόρμα που συγκεντρώνει διάφορες οργανώσεις που συζητούν θέματα αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού και πολλών άλλων συνεργασίων συνεργαζόμαστε λοιπόν για να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινά σημεία τα οποία να οδηγούν σε μια κοινή μορφή διακρίσεων. Έχουμε δημιουργήσει αυτή την πλατφόρμα η οποία μας βοήθησε να προτείνουμε καλές οδηγίες βάσει αυτού του άρθρου 13. Εάν λοιπόν κοιτάξτε την κατάσταση στην Αυστρία προσφάτως με τον κύριο Χάιντερ μας υποκίνησε να δουλέψουμε και ούτως ή άλλως δεν έχουμε ε, τελειώσει ε, την, ε, τα μέτρα ενάντια στις διακρίσεις. Τώρα λοιπόν πρέπει να δούμε σχετικά με την θέση, με την ισότητα των φύλων στον χώρο της εργασίας τι θα πει το Συμβούλιο. Ε, δεν ξέρω λοιπόν αν ε, είναι ε, το Ινστιτούτο αυτό ένα, μια περιττή πολυτέλεια διότι θα μπορούσε να έχει ενσωματωθεί σε έναν άλλο οργανισμό. Καλύτερο θα ήταν λοιπόν ο οργανισμός αυτός να μην συνδυάζει τη χειραφέτηση και με τις πολιτικές ισότητος. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με θέματα ισότητος αλλά και με άλλους, άλλες αιτίες διακρίσεων όπως ε, είναι οι αναπηρίες διότι ό,τι έχει σημασία για τους αναπήρους έχει σημασία για ε, όλους και ό,τι έχει σημασία για τους νέους έχει πάλι σημασία για όλους. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι η ισότητα των φύλων είναι απλώς μία προοπτική για να επιτύχουμε ίση μεταχείριση για όλους. Ανακεφαλαιώνοντας έχω δεκαετίες εμπειρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη για την εργασία η οποία είναι σημαντική σε αυτή την Επιτροπή και τρίτον έχω ένα όραμα το οποίο να ακολουθεί την εργασία που έχετε κάνει στον τομέα αυτό. Ελπίζω ότι θα μου επιτρέψετε να συμβάλλω στο Ινστιτούτο διότι αξίζει. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Παρακαλώ, δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις από τα μέλη της Επιτροπής μετά από αυτή την παρουσίαση. Υπάρχουν ερωτήσεις. Ε, σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που σας συναντώ. Ε, ήρθατε πολλές φορές με την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα για το θέμα της ισότητας των δύο φύλων και θα ήθελα να σας θέσω το εξής ερώτημα. Αναλαμβάνονται διαρκώς πρωτοβουλίες ε, σε αυτό το τομέα και ποτέ δεν επαρκούν. Είπατε και εσείς οι ίδια ότι οι πόροι του Ινστιτούτου θα είναι περιορισμένοι. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή λόγω οικονομικής κρίσης. Ε, έχουν δοθεί ε, πολλοί πόροι στις τράπεζες ε, δισεκατομμύρια, αλλά όταν μιλάμε για τους πόρους, για την αναβάθμιση της κατάστασης της ζωής των γυναικών, ποτέ δεν γίνονται δεκτές οι προτάσεις με την πρόφαση ότι δεν υπάρχουν αρκετά κονδύλια. Ε, σε αυτό το φόρουμ των εμπειρογνωμών πώς ακριβώς θα αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση. Ε, ποιες θα είναι οι συμβουλές σας προς, ε, τους, προς τη διεύθυνση του Ινστιτούτου. Σας ευχαριστούμε. Ακούμε την απάντησή σας, παρακαλούμε. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, ναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα ε, που θα πρέπει να στοχεύσει τη δράση του ε, το Ινστιτούτο. Θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια αντίστοιχη γραμμή όπως αυτή του Ινστιτούτου με το οποίο συνεργάζομαι στην Ολλανδία. Θα μπορούσαμε σε μια άλλη κλίμακα να ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική αλλά δεν μπορούμε να επανεφεύγουμε τον τροχό ούτε το χρόνο έχουμε ούτε την απαιτούμενη ενέργεια. Ήδη έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, πάρα πολλές έρευνες. Το σημαντικό είναι να χρησιμοποιήσουμε τα πορίσματα των ερευνών, να τα δημοσιεύσουμε, να τα κοινοποιήσουμε και να ε, προσθέσουμε και τις δικές μας γνώσεις, τη δική μας τεχνογνωσία. Δεν πρέπει πάντοτε να προσπαθούμε να ε, κυνηγάμε όλοι τους ίδιους στόχους, θα πρέπει να αναλαμβάνουμε και πρωτοβουλίες. Όταν μιλάμε για μερική απασχόληση, για διαμητρότητας, νομίζω ότι δεν πρέπει να θέτουμε έτσι το ερώτημα. Είναι ζήτημα οργάνωσης των εργασιών μας για να υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε κι άλλες ε, δύο ερωτήσεις, μία από μένα και μία από την κυρία Μπάουερ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για την σημασία του gender mainstreaming, ε, τονίσατε αυτό το θέμα στην παρουσίασή σας ε, και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι για την ε, υλοποίηση. Όλοι μιλάνε για το gender mainstreaming, για το gender budgeting, αλλά πώς θα ε, τα καταφέρουμε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα. Ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι διακριτικής μεταχείρισης. πέρα ε, από το φύλλο έχουμε την ηλικία, τις αναπηρίες, ε, υπάρχει μια σειρά λόγων διακριτικής μεταχείρισης και σας ε, ερωτώ. Το Ινστιτούτο Ισότητας των Ευκαιριών με ποιο τρόπο θα μπορέσει να συνεργαστεί με τα λοιπά Ινστιτούτα που ασχολούνται με τους υπόλοιπους λόγους διακριτικής μεταχείρισης πέραν του φύλλου. Κοιτάξτε. Ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα του gender budgeting και του gender mainstreaming. Ε, οφείλουμε να ριοθετήσουμε το πρόβλημα του, που σχετίζεται με το gender mainstreaming για να βρούμε τη λύση. Ε, το θέμα είναι πάντοτε να ακολουθούμε μία ε, διπλή πολιτική για να έχουμε αποτελέσματα. Για τους κανονικούς εφακέλους πρέπει να συνεχίσουμε να επιμένουμε στο θέμα της ισότητας και ε, από την άλλη πλευρά θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτως ώστε οι πολιτικές να είναι πολυδιάστατες. Για το gender budgeting Γι' αυτό το θέμα πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να υπάρχει η πραγματική βούληση. Ε, ανέκαθεν εμείς στην Ολλανδία ζητάμε ε, φορολογικές προσαρμογές. Ε, έχουμε υπερασπιστεί αυτή την αρχή. Το Υπουργείο Οικονομικών τελικά ε, δέχτηκε να εξετάσει ε, διάφορες φορολογικές προσαρμογές. Και έτσι δίνουμε το καλό παράδειγμα και αυτό πάντοτε είναι χρήσιμο. Τώρα, πώς ε, να εξασφαλίσουμε μια αγαστή συνεργασία ανάμεσα στο Ινστιτούτο της Ισότητας των Δύο Φύλων και το Ινστιτούτο στη Βιέννη. Παραδείγματος χάρη. Ας πάρουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για ε, τις αναπηρίες. ξέρετε, η χειραφέτηση των γυναικών ακολουθεί μια παράλληλη πορεία με την ανεξαρτοποίηση ε, των ατόμων με αναπηρίες. Δηλαδή μπορούν να αντλήσουν διδάγματα από τη δράση που έχουμε εμείς στον τομέα της ισότητας των δύο φύλων. μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, την τεχνογνωσία μας για να φέρουν, ε, επιφέρουν ε, αλλαγές και στο δικό τους τομέα. Εγώ βλέπω ότι συμβαίνει αυτό στην Ολλανδία με τα άτομα με ειδικές ανάγκες, με μια οδηγία που έχει ένα, ένα νομοσχέδιο που έχει εγκριθεί για την πρόσβαση των αναπήρων, παραδείγματος χάρη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να μάθουμε ημένα από τους ΔΕΝ μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και τις καλύτερες πρακτικές για να σημειωθούν γρήγορα εξελίξεις. Έχουμε άλλες τρεις ερωτήσεις να ακούσουμε πριν ολοκληρώσουμε το σημείο αυτό. Η κυρία ε, Μπάουερ, η κυρία Κορνέλη και η κυρία Κλάς. Κυρία Μπάουερ, αρχίζει παρακαλώ. Ευχαριστώ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, πρόκειτο για μία έκθεση. Ε, ήταν η δική μου η έκθεση και δεν μπορούσα να μην είμαι παρούσα. Αυτό που είπατε είναι πολύ ενδιαφέρον ότι χρειαζόμαστε νέες πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα από αυτού, ιδίω από μία συνάδελφο και θα μπορούσα να πω και αντίζηλό σα. ρώτησα τι θα έπρεπε να μας απασχολήσει πρώτα, να ψάξουμε νέες στρατηγικές, να επιζητήσουμε νέα νομοθεσία ή θα έπρεπε να κοιτάξουμε μέχρι ποιου σημείου ισχύουν και εφαρμόζονται οι νομοθεσίες οι οποίες υφίστανται. Δηλαδή πόσο νομότυπη είναι η διαδικασία, τι θεωρείτε εσείς σαν προτεραιότητα. Δεν θέλω να πω ότι το ένα θέμα είναι πιο επουσιώδης από το άλλο, αλλά εάν καταρτίζατε προτεραιότητες, τι θεωρείτε ότι είναι προτεραιότητα για τη δουλειά του Ινστιτούτου. Ε, ειλικρινά Νομίζω ότι χρειαζόμαστε ορισμένες ε, ε, νέες νομοθεσίες δεν πρέπει δηλαδή να επιμείνουμε, μάλλον θα έπρεπε να δούμε τι γίνεται παραδείγματο χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για να ε, γίνει γνωστή η νομοθεσία, να διαδοθεί η υιοθέτηση της ε, νομοθεσίας είναι κάτι βασικό για το Ινστιτούτο. Βεβαίως όπως είπατε πρέπει να βρούμε νέες στρατηγικές και αυτό είναι βασικό διότι και 30 ή και 50 χρόνια νομοθετούμε και ε, διατυπώνουμε πολιτικές με τον ίδιο τρόπο. Ξέρετε ότι έχουμε προχωρήσει αλλά δεν έχουμε λύσει όλα τα θέματα ακόμη. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πραγματικά ε, προστιθέμενη αξία εάν μπορούσαμε εδώ να έχουμε ε, ένα αποτέλεσμα. Η κυρία Κορνίλσεν. Uh, Είπατε απαντώντας σε μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις ότι η οργάνωσή σας ε, μοιάζει με το Ινστιτούτο Ισότητας ε, των Δύο Ευκαιριών ε, και μου τράβηξε αυτό την προσοχή. Μπορείτε να μας μιλήσετε για τις ομοιότητες ανάμεσα στα δύο Ινστιτούτα. Yes. Um, well, what, we in, κοιτάξτε, ναι. Στο Ινστιτούτο με το οποίο συνεργάζομαι ε, κοιτάζουμε τι μελέτες έχουν γίνει από άλλα Ινστιτούτα και τις προσαρμόζουμε για τις μη ή για ε, τις ε, κρατικές αρχές, ε, για χρήση δηλαδή από τις μη καπαόμικρον και από τις κρατικές αρχές. Η κυβέρνηση ενίοτε μας ζητάει συμβουλές για θέματα όπως η άδεια μητρότητας, ε, η φροντίδα των παιδιών ε, και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ε, δίνουμε συμβουλές ή να βοηθάμε παραδείγματος χάρη τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αν θέλουν βέβαια να επιχειρήσουν κάτι δεν είναι σημαντικό τι πιστεύουμε εμείς απλά τις βοηθάμε να έρθουν σε επαφή με την κυβέρνηση. Τις με κυβερνητικέ οργανώσει, αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Σας ευχαριστούμε. Μία τελευταία ερώτηση από την κυρία Κλάς. Ευχαριστώ. Στην ε, εισαγωγή σας αναφερθήκατε στο βιογραφικό σας και είπατε ότι αυτό ήταν ε, συνοπτικό. Πρέπει όμως να σας πω ότι είναι πολύ εκτενές και διάφορα πράγματα δεν τα καταλαβαίνω και γι' αυτό επανέρχομαι. Καταρχήν όμως όταν λέτε μεταξύ άλλων ότι έχετε αναλάβει πολλά καθήκοντα με τα οποία συνεχίζετε θεωρείτε ότι δεν γίνετε εμπειρογνώμων στο Ινστιτούτο το αυτό θα μπορέσετε στο μέλλον να συνεχίσετε την εξάσκηση αυτών των καθηκόντων. Μπορεί να υπάρχει ε, σύγκρουση και ίσως θα έπρεπε να σχολιάσετε και αυτό. Είπατε ότι είσαστε πολιτικός και ε, μέλος της Επιτροπής για την ε, ε, ε, ε, για την οικειοθελή ευθανασία και γενικώ νομίζω ότι πρέπει να μας σχολιάσετε λιγάκι για να δούμε ακριβώς τι κάνετε. Ευχαριστούμε κυρία Κλά, σας ακούμε για όλα, όλες τις θέσεις που είχα στο παρελθόν. Κοιτάξτε, εάν ε, ρωτήστε κάτι που είναι ήδη, ε, κάποιον ε, που είναι ήδη αποσχολημένος θα σας πει ναι, ναι, ναι, μπορώ να το αναλάβω γιατί δεν είναι τόσο σημαντικό αν προσθέσετε και άλλη μια ώρα δουλειά αν ούτως ή άλλως δουλεύετε μέχρι τα μεσάνυχτα, για μένα αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. για τους ε, αγώνες ομοφιλοφίλων Gay Games κάθε χρόνο ε, διοργανώνεται ε, μια μεγάλη εκδήλωση. Το 1998 είχαμε τα Gay Games στην Ολλανδία. Και βοηθήσαμε τις χώρες για την οργάνωση. Τους πρόσφερα δηλαδή την τεχνογνωσία μου για την ευθανασία. Το πιο Η πιο σημαντική συνεισφορά μου είναι να τους βοηθήσουν να έρθουν σε επαφή με διάφορες πολιτικές ομάδες, με διάφορα κόμματα, γιατί φοβούνται λίγο και εγώ ε, τηλεφωνώ εκ μέρους τους, ώστε να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμά τους. Αυτά. Σας ευχαριστούμε εξ ονόματος της Επιτροπής σας ευχαριστώ θερμά για την ε, παρουσίασή σας. Ε, ήταν σαφείς οι απαντήσεις που μας ε, δώσατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν και καλή επιτυχία για το μέλλον. Συνάδελφοι, έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πώς ε, να παρεμποδίσουμε, να εξαλείψουμε τη βία κατά των γυναικών. Είναι ένα θέμα που ήδη συζητήσαμε επί μακρόν σήμερα με τους προσκεκλημένους μας. Την 1η Σεπτεμβρίου αποφάσισαν οι συντονιστές ότι η Επιτροπή μας θα υπέβαλε μια προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή για το Συμβούλιο για τη βία κατά των γυναικών. Αποφασίσαμε επίσης να εκδώσουμε ένα σχετικό ψήφισμα διότι Έχουμε την ε, Διεθνή ημέρα ε, καταπολέμησης της βίας κατά των ε, γυναίκων. Είναι η δέκα τέτοια μέρα. Και σήμερα καλούμαστε να αποφασίσουμε για την προφορική ερώτηση. Το ψήφισμα θα το δούμε μεταγενέστερα. Σήμερα χρειάζεται μία απόφαση μόνο για τις προφορικές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Όλα τα μέλη της Επιτροπής έχουν ε, δραστηριοποιηθεί ε, ήδη ε, και έχουν εργαστεί για αυτές τις προφεωρικές ερωτήσεις και συμμετείχαν με ιδιαίτερα ενεργό τρόπο για να συντάξουμε αυτές τις προφορικές ερωτήσεις. Απλά ήθελα να διευκρινίσω και κάποια πράγματα για το ψήφισμα Οι μεταφράσεις θα είναι διαθέσιμες από τις 5 Οκτωβρίου και μετά. Μετά, όλοι οι συνάδελφοι θα μπορέσουν να υποβάλουν τροπολογίες για το ψήφισμα μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Και μετά θα ακολουθήσουμε τη συνήθεια διαδικασία για τα ψηφίσματα. Στις 4 Νοεμβρίου θα ληφθεί απόφαση στην Επιτροπή μας ε, και στην ε, ε, δεύτερη Ολομέλεια και του Νοεμβρίου θα υποβληθεί η ερώτηση. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό που ελήφθη η απόφαση ναι, για να υποβάλουμε τις προφορικές ερωτήσεις και αυτός είναι και ένας λόγος που αποφασίσαμε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα είναι η διεθνή ημέρα κατά της βίας, ε, κατά των γυναικών και αυτό είναι το βασικό έρισμα για τις ερωτήσεις και το ψήφισμα, βασικότερος λόγος είναι ότι συμφωνούμε όλοι μας πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρεμποδίσουμε και να σταματήσουμε ε, αυτή την απαράδεκτη βία που πλήττει τόσες πολλές ε, γυναίκες. Ε, δεν μιλάμε μόνο για την, το ότι πλήττει την υγεία τους, μιλάμε για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική, στην οικονομική ζωή, σε όλους τους τομείς ε, δραστηριότητα στην κοινωνία μας. Είναι επίγον, είναι σημαντικό ε, για την Επιτροπή μας να εντατικοποιήσει τις εργασίες που έχει αναλάβει στον τομέα αυτό γιατί φέρουμε μεγάλη ευθύνη για τις γυναίκες και στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές ε, του κόσμου. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε στον τομέα αυτό. Εν συντομία θα ήθελα να σας πω ότι είναι εξαιρετικά επίκαιρο το θέμα διότι η Σουηδική Προεδρία προετοίμασε το επωνομαζόμενο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, για την ασφάλεια, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη και βλέπουμε ένα σαφή ε, δεσμό με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων των γυναικών να ζουν χωρίς τη βία. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στα δύο και μιλάμε για την δικαιοσύνη, ε, για τα δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης και Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία και χαίρομαι που τα μέλη της Επιτροπής ε, ανέλαβαν αυτή την πρωτοβουλία για την υποβολή των προφορικών ερωτήσεων και την ε, εκπόνηση του ψηφίσματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να δω πως υπάρχουν ε, παρατηρήσεις. Η κυρία Μαντέιρα έχει ήδη ζητήσει το λόγο και στη συνέχεια η κυρία Γκαρσία Πέρες. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την καθυστέρηση με την οποία ήρθα σήμερα. Ευτυχώς σήμερα είναι πολύ σημαντική ε, μέρα για την Επιτροπή Προεπιλογισμού. Ζητώ ε, συγγνώμη λοιπόν. Και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτείτε και τις δύο τροπολογίες μου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλήσω σήμερα και να παρέμβω ως ε, σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ για τις δύο προφορικές ερωτήσεις, δεδομένες και τη σημασίας που έχει ε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ασχοληθούν με αυτό το θέμα της βίας κατά των γυναικών. Εγώ ζήτησα αλλαγή του αρχικού κειμένου της προφορικής ερώτησης ε, που απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο συγκεκριμένα εκεί που αναφερόμαστε σε ένα ε, γύρο τραπέζις ε, εμπειρογνωμόνων σε υψηλό επίπεδο. Εγώ ήθελα να μιλάμε για μια ειδική διάσκεψη, να μην υπάρχει μια κάποια χρονική αναφορά και επίσης ήθελα να προτείνω ότι πρέπει να αναφέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη οι εκπρόσωποι πολιτικών οργανώσεων, ε, της κοινωνίας των πολιτών, των ε, θεσμικών και κοινωνικών οργανώσεων. Και επιπλέον, και ολοκληρώνω με αυτό, πρότεινα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε και ποιος ε, πρέπει να είναι σκοπός αυτής της παρέμβασης που είναι να δώσουμε μια μεγαλύτερη όθεση για την ανάπτυξη πιο συνεκτικών πολιτικών ε, για την ε, βία ε, κατά των γυναικών. Να σας ευχαριστώ λοιπόν για άλλη μια φορά κυρία Πρόεδρε που δεχτήκατε τις τροπολογίες μου και ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρθία Πέρες παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε συμφωνώ με την ανάγκη το Κοινοβούλιο να εκφράσει την άποψή της ε, για μια αλήθεια, μια πραγματικότητα σαν αυτή που, ε, της βίας κατά των γυναικών ε, την οποία τη βλέπουμε σε όλα τα πολιτικά επίπεδα για την εξάλληψη αυτής της κοινωνικής μάστιγας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα για ένα κοινό ψήφισμα για να ακουστεί ε, βροντερά η φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτό το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για να μπορέσουμε να τροποποιήσουμε ίσως το κείμενο της προφορικής ερώτησης, διότι διαπίστωσα ότι υπάρχει μια δήλωση στην προφορική ερώτηση, η οποία θεωρώ ότι δεν είναι η πλέον κατάλληλη λέει ότι κανένα από τα κράτη-μέλη δεν έχουν ε, επιτυχία στην επίλυση αυτής της κατάστασης δεν ε, υπάρχει καμία αμφιβολία ότι προκειμένου να επιληθεί ένα πρόβλημα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι υφίσταται. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να ε, κλείνουμε τα αυτιά μας και να λέμε ότι όλα όσα γίνονται είναι καλά και επιτυγχάνουμε όλα τα κατάλληλα αποτελέσματα. Αλλά από την άλλη δεν μπορούμε και να πούμε ότι δεν επιτυγχάνεται τίποτα διότι ε, θεωρώ ότι σε νομοθετικό επίπεδο προωθούνται μέτρα τα οποία είναι σημαντικά, τα οποία ε, μπορεί ίσως ε, βραχυπρόθεσμα να μην βελτιώνουν τα στατιστικά της στοιχεία που έχουμε για θύματα κακομεταχείρισης, αλλά μπορούν να επιτύχουν κάποιες μακροπρόθεσμες πολιτικές, όπως για παράδειγμα η παιδεία, η πρόληψη, η επιμόρφωση του προσωπικού που εργάζεται σε τέτοια θέματα. Ε, αυτά όλα δεν είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να έχουν αποτελέσματα εν μία νυχτή. Θα πρέπει να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν κάποια θετικά βήματα. Είναι πολιτικές μακροπρόθεσμες, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πόσο αποτελεσματικές είναι και θα ήθελα να ζητήσω, ε, δεν ξέρω, ή να διαγράψουμε αυτή τη φράση. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συνειδητοποιούμε ποια είναι η πραγματικότητα, αλλά θα πρέπει λίγο να εμπιστευτούμε τα μέτρα τα οποία προωθούνται, τα οποία ε, φρονώ ότι είναι θετικά. Σας ευχαριστούμε κυρία Γκασία Πέρες. Ε, να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο ε, σε σχέση με αυτά που είπατε. Δηλαδή, ότι πρέπει να δούμε και ποιο ποσοστό επιτυχίας είχαν τα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, κατά τη γνώμη μου θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι απαραίτητο να, να συμμετάσχει κανείς στην προφορική ερώτηση. Θα δούμε τι πιστεύουν και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, αλλά μπορούμε και να τη βγάλουμε αυτή ε, την πρόταση αν δημιουργείται παρανόηση. Ε, η κυρία Σινκλέρ και η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας συγχαίρω ε, και εγώ ε, παθιάζομαι για αυτό το ζήτημα και έχω δουλέψει πολύ στην εκλογική μου περιφέρεια για να το προωθήσω. Εγώ ε, θα ήθελα να υποστηρίξουμε τα κράτη-μελή για να εκπονήσουν εθνικά σχέδια δράσης. Αυτή η πρόταση πρέπει να παραμείνει μέσα στο ψήφισμα. Ε, ε, ε, με την εντολή που μου έχει ανατεθεί φυσικά δεν θα αντιταχθώ σε μια κοινοτική νομοθεσία και αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε αυτήν την ημέρα το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα θα σας υποστηρίξω ε, να ευχαριστήσω πολύ την ε, Πρόεδρο που ε, υπέβαλε αυτή την πολύ σημαντική προφορική ερώτηση που θα δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επισημάνει αυτό το θέμα και να δείξει και τι ακριβώς κάνει σε τόσες πολλές γυναίκες που περιμένουν απαντήσεις από εμά. Ήθελα να προτείνω μία μικρή διόρθωση η οποία είναι σημαντική για μένα στο προήμιο όταν λέτε ότι η βία κατά των γενικών δεν είναι μόνο θέμα δημόσιας υγείας αλλά και θέμα ανισότητας, αίτιο ανισότητας εγώ θα ήθελα να προσταθεί και προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου. Δεν είναι μόνο θέμα ανισότητας, αλλά είναι μια σοβαρή προσβολή της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου και είναι από τα θέματα τα οποία βρίσκονται στα χάρτα των αξιών μας. Και Διερωτέμαι. μια πάρα πολύ μικρή πρόταση, αλλά νομίζω ότι τα απαντήσατε κι εσείς και είπατε ότι όταν γίνεται η προφορική ερώτηση, αυτός που απαντάει είναι αυτός που θα διευκρινίσει. Αυτό που θα ήθελα ίσως να προκύψει λίγο περισσότερο στη συζήτηση είναι ένα θέμα το οποίο εμείς ε, σήμερα ως γυναίκες δεν έχουμε εξετάσει επαρκώς, που είναι το θέμα του τι ακριβώς ε, πρέπει να κάνουμε ως προς την ε, κατάχρηση της εικόνας και του πολύ σοβαρού ε, τρόπου ε, με τη μορφή καρικατούρας ε, ή κάποιες φορές προσβλητική μορφή με την οποία παρουσιάζονται οι γυναίκες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Νομίζω ότι και η νέα οδηγία για την τηλεόραση χωρίς σύνορα που περιλαμβάνει και κάποιους κώδικες διοντολογίας ε, δεν ε, γίνεται σεβαστή στο ελάχιστο. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία έκκληση πολύ πιο στεναρή στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το αφήσουμε και στις προφορικές παρεμβάσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει και στη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Απλά ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που μας είπε η κυρία Κώστα. Συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, αυτή η ερώτηση γιατί υπάρχει και στο ψήφισμα αλλά δεν υπάρχει αυτό το σημείο στην προφορική ερώτηση, γιατί πρέπει να την περιορίσουμε στο μέγεθό τη και ούτω ή άλλω μπορούμε να το αναφέρουμε όταν θα γίνει συζήτηση για το ψήφισμα. Ελπίζω να συμφωνούν εκεί οι συνάδελφοι ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ακουστεί και αυτή η άποψη. Λοιπόν, νομίζω μπορούμε να αποφασίσουμε τώρα για, την προφο... για τις ε, προφορικές ερωτήσεις. Δέχεστε, εγκρίνετε την προφορική ερώτηση με την προφορική τροπολογία που έκανε η κυρία Γκαρσία Πέρες που διευκρινίζει ότι θα διαγράψουμε αυτή την πρόταση σχετικά με την επιτυχία που έχουν σημειώσει τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πολύ ωραία. Δεν χρειάζεται καν να ψηφίσουμε. Ομόφωνα εγκρίνουμε αυτές τις δύο προφορικές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συνεδρία. Η κυρία Μπάουερ μας ζήτησε το λόγο, παρακαλώ. Συγγνώμη. Ε, έχω επίγνωστο ότι αργοπόρησα, δεν ζήτησα γερός το λόγο. Εγώ υποστηρίζω αυτή την πρόταση που κάνατε για να διαγραφεί αυτή η αράδα που αναφέρεται στην επιτυχία ή έλλειψη επιτυχία στην αντιμετώπιση του ζήτηματο από τα κράτη-μέλη. Στο βαθμό που είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα, χρειάζεται κοινή δράση. Πώς έπρεπε να το πούμε κάπως έτσι. Και θα ήθελα να συμπεριληφθεί ε, και αυτό το κομματάκι για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την αξιοπρέπεια των γυναικών. Ε, νομίζω είναι απαραίτητο να το αναφέρουμε. Ε, δεν είναι και πολύ σημαντική η τροπολογία μου. Ναι, ευχαριστούμε κύρια Μπάουερ. Ξαναλέω ότι ε, τα περί αξιοπρέπειας υπάρχουν στο ψήφισμα. Ε, θα γίνει συζήτηση για το ψήφισμα και όλοι οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν τροπολογίες και ε, έτσι θα γίνει διεξοδική συζήτηση για αυτό το θέμα. Τώρα, για την προφορική ερώτηση πρέπει να αποφασίσουμε σήμερα και από ό,τι κατάλαβα συμφωνούν οι συναδελφοί να εγκριθούν αυτές οι προφορικές ερωτήσεις με την προφορική τροπολογία της κυρίας Γκαρσία Περές. Σωστά εννοήσα, εγκρίναμε τις ε, προφορικές ερωτήσεις. Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ τη γραμματεία. Ευχαριστώ όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτό το ενδιαφέρον απόγευμα. Αύριο οι συντονιστές θα αποφασίσουν ε, για τους υποψηφίους για το Φόρουμ Εμπειρογνωμόνων. Σας ευχαριστώ και ε, θα ε,